Παρακαλώ καθίστε για να ξεκινήσουμε, έχουμε ήδη καθυστερήσει. Οι εργασίες μας σήμερα είναι πολύ φορτωμένες. Δεν χρειάζεται να δοκιμάσουμε τις κάρτες μας στο ηλεκτρονικό σύστημα. Απλά μόλις την τοποθετήσετε στο μηχάνημα τότε θα εμφανιστεί το όνομά σας. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε συνδεδεμένοι και μπορούμε να ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες στο πρώτο σημείο της μεσίας διατάξεως που αφορά την έκθεση Oman Royten σχετικά με την έκθεση προόδου της Τουρκίας. Περνάμε με την τροπολογία 9, παράγραφος 1, ψήφι υπέρ. Συγγνώμη, συγγνώμη. Τροπολογία 28, υπέρ. Παρακαλώ, διανατάσσεως της χειρός. Κατά. Απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο επί της 28, ωραία. Ψηφίζουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας, αποτέλεσμα. 30 ψήφι κατά, 20 κατά. Μήπως κάποιο μηχάνημα ηλεκτρονικό δεν λειτουργήσε. Λοιπόν, δύο, τρεις ψήφοι κατά. Ε, πρόεδρος, λοιπόν, Το τελικό αποτέλεσμα είναι 32 ψήφοι κατά και 20 υπέρ. Απορρίπτεται τροπολογία 29. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ κατά απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 32. Ψήφι υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 33 υπέρ κατά απορρίπτεται. 34 υπέρ όχι συγγνώμη έχει καταπέσει 34 καλύπτεται από το Σύμβασμα περνάμε στο Σύμβασμα υπάρχει μόνο δύο ψήφοι υπέρ κατά <clears throat> εγκρίνεται 35 36, 37 και 38 καλύπτονται το συμβασμό 2. Περνάμε συμβασμό 3. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 48. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 49 υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 50 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 51 ψήφι υπέρ ψήφι κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Δεκτός. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 και 60 καταπίπτουν. Προφορική τροπολογία της εισηγήτριας. Η κυρία Φιλότρο έχει το λόγο. Παρακαλώ. Εδώ έχουμε και την προφορική τροπολογία της εισηγήτριας που λέει ότι ιδιαίτερα για την απόφαση περί εφαρμογής, περί ανέρεσης παρακύρωσης ε, νομοθεσίας από το Σταματικό Δικαστήριο και προτείνει, ε, συνιστά την ε, πρόοδο σε μια σταματική μεταρρύθμιση ως προσθήκη με την προφορική μου τροπολογία, ως προς την τροπολογία της συγκεκριτρίας. Η συγκέντρια δέχεται αυτή την πρόταση. Ναι, Πρόεδρε, συμφωνώ. Αλλά έγινε σχετική συζήτηση χτες για το θέμα αυτό και απάντησα προς την κυρία Φλότρου. Χαίρομαι που άλλαξε τώρα την προφορική της τροπολογία. Λοιπόν, ψηφίζουμε την τροπολογία με την τροποποίηση της προφορικής τροπολογίας ψηφί υπέρ κατά 61 υπέρ κατά απορρίπτεται 62 υπέρ κατά απορρίπτεται. Δεν ε, αναφέρω τις ε, αποχές, ε, απλά για να επιταχύνουν τη διαδικασία υπέρ. 63 τροπολογία υπέρ. Κατά. Δεκτή. Διαμαρτυρίες. Απορρίφθηκε, εντάξει. 64. Εντάξει, ελέγχουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 63. Πέρα ψηφοφορίες. Τελικό αποτέλεσμα. 44 συν 1, 45 ψήφοι κατά, 20 υπέρ, απορρίπτεται όπως πολύ σωστά είπατε. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. 65. λάμπστορφ Εδώ έχουμε μια προφορική τροπολογία που τη βλέπετε στο έγγραφο. Ψήφι υπέρ. Κατά. Δεκτή. 66 υπέρ. Κατά. Ας επαληθεύσουμε. Ψηφίζουμε επί της 66. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία επί της 66. Έληξε ψηφοφορία. Τελικό αποτέλεσμα. 26 ψήφοι κατά, 34 υπέρ. Συν ε, ε, μία ψήφος κατά που δεν μπορεί να εκφραστεί ηλεκτρονικά, 27 λοιπόν. Άρα καταπίπτει, περνάμε στην 68 <clears throat> υπέρ. Κατά, απορρίπτεται. 69 υπέρ. Κατά, απορρίπτεται. 70 προφορική τροπολογία τι βλέπετε στο κείμενο. Ψήφι Κατά. Δεκτή. 71. Ψήφι Κατά. Απορρίπτεται. 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 73. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 74. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 75. Υπέρ. Κατά. Δεν είμαι σίγουρος για το αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικός. 75. Άρχιτε ψηφοφορία. 75. Έληξη ψηφοφορία. Δύο ψήφοι αθρίζονται διότι το μηχάνημα δεν λειτουργήσε. 35 ψήφοι υπέρ, 35 ψήφοι κατά. Απορρίπτεται λόγω ισοψηφίας. Πρόεδρε, δεν έχω ε, κάρτα ψηφοφορία, αλλά ήθελα να ψηφίσω υπέρ. Va bene, allora con 36 a 35 τότε 36-35 εγκρίνεται. 60, 76 καταπίπτει, 77 ψήφι Κατά. Λοιπόν, 77 θα ψηφίσουμε σου. Άρχιτε ψηφοφορία. Έληξε ψηφοφορία. Αποτέλεσμα. Μα τότε δεν ψηφίσετε, δεν σηκώνετε το χέρι σας, 56 ψήφοι κατά και 10 ψήφοι υπέρ. Απορρίπτεται. 78, πανόρτον, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 79 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 80 υπέρ. Κατά. Καλύτερα να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 80. Έληξη ψηφοφορία. Τελικό αποτέλεσμα. 35 πέντε ψηφιπέ, τριάντα κατά. εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 83. <clears throat> Προφορική τροπολογία, το βλέπετε στο κείμενό σας. Ψήφι υπέρ. Κατά. Δεκτή. 84. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 85 υπέρ κατά απορρίπτεται 86 υπέρ κατά απορρίπτεται συμβαστική 6 υπέρ κατά δεκτή περνάμε στην 95 διότι οι προηγούμενε καταπίπτουν υπέρ 95 κατά απορρίπτεται 96 υπέρ κατά απορρίπτεται 97 όχι όχι καλύπτεται από το συμβασμό συμβασμός 7 ψήφι υπέρ κατά δεκτός 100 ψηφιπέρ κατά δεκτή 101 υπέρ κατά απορρίπτεται 102 θα ψηφίσουμε μόνο το τελικό κομμάτι της τροπολογίας ψήφι υπέρ. Κατά. Δεκτή. 103 τροπολογία υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 104 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 105 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 106 υπέρ κατά απορρίπτεται 107 <clears throat> υπέρ κατά απορρίπτεται 108 υπέρ κατά απορρίπτεται 109 υπέρ κατά απορρίπτεται 110 του υπέρ κατά απορρίπτεται 111 υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβαστική 8 της εισηγήτρια ψήφι κατά δεκτή. Καταπίπτουν οι πιστροπολογίες, φτάνουμε στα 115 υπέρ. Κατά απορρίπτεται 116 προφορική τροπολογία την έχετε στο έγγραφό σας ψηφιπέρ κατά δεκτή 116, 117, 118 καταπίπτουν και 119 περνάμε στην 120 υπέρ, κατά απορρίπτεται 121 υπέρ κατά απορρίπτεται 122 υπέρ κατά απορρίπτεται 123 υπέρ, συγγνώμη, χωριστή ψηφοφορία, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, απορρίπτεται, δεύτερο τμήμα της 123 ψήφι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 124 να ξαπολύσουμε το πρώτο τμήμα του 123, άρα να ψήφουμε το 124, ψήφι υπέρ 124. Κατά. Απορρίπτεται. 125 υπέρ. Κατά. Α επαληθεύσουμε ηλεκτρονικός. Άρχιε η τροπολογία του 125. η ψηφοφορία. Αποτέλεσμα 41 ψήφοι κατά 30 υπέρ. Απορρίπτεται 126 ψήφοι υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται 127 προφορική τροπολογία ψήφοι υπέρ. Κατά δεκτή 128 υπέρ. Κατά Ε, νομίζω πως απορρίφθηκε. Δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία, δεν σηκώνει τα χέρια σας, κάνετε δύσκολη τη ζωή. Εγώ νομίζω ότι απορρίφθηκε. Δεν πέστε 129 υπέρ. Α, για την 128 θέλετε να επαληθεύσουμε. Ωραία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικώς την 128. Έληξε η ψηφοφορία. 45 ψήφοι κατά, 27 υπέρ, απορρίπτεται. Ε, παρακαλώ να συμμετέχετε. 129. Σαλαφράγκα. Πρόεδρε, διαδικαστικό θέμα. Θα ήθελα να επαληθεύσετε πόσοι συμμετέχουν στις ψηφοφορίες από κάθε πολιτική ομάδα γιατί έχουν την εντύπωση ότι ε, ψηφίζουν περισσότερα μέλη από τα μέλη της Επιτροπής. Εντάξει, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά καλύτερα να το επαληθεύσουμε λοιπόν. Να μην ψηφίζουν περισσότερα μέλη. Λοιπόν, η εξήγηση που μου δίνεται από τη γραμματεία είναι η εξή. Υπάρχουν όντως δύο επιπλέον από τη δική μας πολιτική ομάδα, αλλά επειδή η Ρία και ο Μπρόκ δεν έχουν την κάρτα τους, τότε αυτό αντισταθμίζεται με τους δύο επιπλέον. Όπως βλέπετε λοιπόν δεν υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να είναι σωστή η ψηφοφορία, όπως διεξάγεται. Λοιπόν, 129 υπέρ. 129 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 130 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ. <clears throat> Κατά. Δεκτό. Δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 131 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Όχι, ας απαλληθέψουμε. 131. Άρχεται ψηφοφορία. Ηλεκτρονικός. Έληξε η ψηφοφορία. Αναφέρεται ότι το ΕΛΚ έχει επιπλέον δύο ψήφους, διότι φαίνεται ότι άρχισαν να λειτουργούν οι κάρτες των δύο συναδέλφων. Εν πάση έχουμε 38 κατά, 32 υπέρ, γίνονται 38, γίνεται 36, απορρίπτεται ούτως ή άλλως. 132 φλότρουν ε, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Για αυτή η πλειοψηφία, Η αυτη η πλειοψηφια συμβαστικη 9 υπέρ, κατά, δεκτή. Και περνάμε στην 135, προφορική τροπολογία, ψηφιπέρ, κατά, εγκρίνεται 136 υπέρ κατά δεκτή 137 προφορική τροπολογία ψήφι υπέρ κατά δεκτή 138 και 139 είναι ταυτόσιμες ψηφιδείς ψηφίζουμε υπέρ κατά απορρίπτεται 140 υπέρ κατά απορρίπτεται 141 υπέρ κατά απορρίπτεται 142 υπέρ κατά απορρίπτεται 143 υπέρ κατά απορρίπτεται 144 σαλαβράκος ψήφι υπέρ κατά απορρίπτεται 145 υπέρ Κατά. Απορρίπτεται. 146. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Καταπίπτει. Όχι, έχει αποσυρθεί, συγγνώμη, 147, 148. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 149. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 150 Χατζη Γεωργίου υπέρ κατά απορρίπτεται 151 Τριανταφυλλίδης ε, πολύ δύσκολο να προφέρω αυτό το όνομα υπέρ 151 κατά απορρίπτεται 152 <clears throat> υπέρ <clears throat> κατά δεκτή. Συμβαστική 10 της ηγήτριας, ε, χωριστά μέρη. Πρώτο μέρος, υπέρ. Κατά, εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος, υπέρ. Κατά, δεκτό. 153. 154-155 καταπίπτουν. Ναι. Περνάμε στην 156 Χωριστή τη ψηφοφορία. Πρώτο μέρος υπέρ κατά Απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος. Όχι, όχι, συγγνώμη. Καλύπτεται από την τροπολογία 10. Περνάμε στην 157. Ούτε. Ξεχάστε την και αυτήν. Έχει. 58-59 έχουν αποσυρθεί. 160-61 καλύπτονται από το συμβασμό 10. 162 έχει αποσυρθεί, 163... Περνάμε στην 164 λοιπόν. Ψηφίζουμε επ' αυτής. 164 υπέρ. Κατά. Αβέβαιο το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονικός την 164. Άρχεται ψηφοφορία. Έληξε ψηφοφορία. Τελικό αποτέλεσμα. 31 ψήφικα. κατά, 37 υπέρ, εγκρίθηκε. Περνάμε στην 165. Όχι, όχι. 166 έχει αποσυρθεί. Τελικά με το ένα και μετά φτάμε 171 ψήφι πέρα. Κατά απορρίπτεται. 172 Σαλαβράκος υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 173 ε, έχει αποσυρθεί. 174 Χατζη Γεωργίου υπέρ κατά απορρίπτεται 175 υπέρ κατά απορρίπτεται 176 υπέρ κατά απορρίπτεται 177 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συγγνώμη 178 υπέρ κατά απορρίπτεται. Το 79 υπέρ κατά απορρίπτεται. 180 θεοχάρους έχει αποσυρθεί, 181 επίσης έχει αποσυρθεί, 182 ψήφι υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 183 έχει αποσυρθεί, 184 υπέρ κατά εγκρίνεται 185 υπέρ κατά απορρίπτεται 186 υπέρ κατά απορρίπτεται 187 υπέρ κατά απορρίπτεται 188 υπέρ κατά απορρίπτεται 189 υπέρ κατά απορρίπτεται 190 υπέρ κατά Α, ας επαληθεύσουμε 190 ηλεκτρονικά άρχεται ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας υπάρχει Πάνε κάποιο που δεν ψηφίζει, α του προσφέρουμε ένα καφεδάκι. 100, λοιπόν, 38 ψήφι υπέρ, 32 κατά, απορρίφθηκε. Πάμε 191 ψήφι υπέρ, κατά. Αποχέ, απορρίπτεται. 192 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 193 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 194 υπέρ κατά απορρίπτεται 195-196 είναι ταυτόσιμες ψήφι υπέρ κατά απορρίπτεται 197 θέλετε να επαληθεύσετε τι ζητάτε 195-196 που είναι ταυτόσιμες ψηφίζουμε ηλεκτρονικός για να ελέγξουμε το αποτέλεσμα. υπάρχουν πάντα δύο, ένας μάλλον, ένας που δεν ψηφίζει. Ποιος είναι αυτός ο ένας επιτέλους. Λοιπόν, το τελικό αποτέλεσμα. 41 ψήφι κατά, 29 υπέρ. Πρόεδρε, εγώ, εγώ δεν ψηφίζω. Δεν έχω το, την κάρτα μου μαζί, γι' αυτό δεν ψηφίζω. Αν δεν έχετε την κάρτα, λοιπόν, αυτό δεν φαίνεται ότι παρίσταστε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Υπάρχει κάποιο το οποίο η κάρτα λειτουργεί, την έχει βάλει στο μηχάνημα, αλλά δεν πατάει το κουμπάκι. Μυστήριο αυτό. 197. Ψήφι πέρα. <clears throat> Κατά. Εκατόν ενενήντα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για να επαληθεύσουμε. Έληξε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τελικό αποτέλεσμα. 29 ψήφοι υπέρ, 41 ψήφοι κατά. Παρακαλώ να συμμετέχετε, να σηκώνετε τα χέρια σας, διότι καθυστερούμε έτσι. 198, καζάκ, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 199, Παπαδόπουλου υπέρ κατά απορρίπτεται 200 υπέρ κατά απορρίπτεται 201 υπέρ κατά απορρίπτεται 202 υπέρ κατά Απορρίπτεται. 203 υπέρ κατά απορρίπτεται 204-206 είναι ταυτόσιμες. Καπαδοπούλου Τριανταφυλλίδης. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 205 Χατζηγεωργίου. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 207 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 208 υπέρ κατά απορρίπτεται 209 υπέρ κατά απορρίπτεται 210 για να, για να κουδάκεις υπέρ κατά απορρίπτεται 211 υπέρ κατά απορρίπτεται 212 μαυρονικόλας υπέρ κατά απορρίπτεται 203 κοπά υπέρ κατά απορρίπτεται 214. Όχι, α, κατα, καταπίπτει. Γιατί η συμβεστική πέντε είναι δεκτή. 215 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 216, 217, 18, 19. Τι κοπέρτη del compromesso 9, Και φτάνουμε εσύ στο 221. Το 221 τροπολογία ΥΠΕΡ, Κατά. Απορρίπτεται. 222 ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 223 Σαλαβράκος. Καταπίπτει. 224 όχι. 225 περνάμε. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 226 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 227 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 228 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 229 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 230 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 231 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 232 υπέρ κατά απορρίπτεται 233 <clears throat> υπέρ κατά απορρίπτεται 234 υπέρ κατά απορρίπτεται 235 και 236 είναι ταυτόσιμες <clears throat> υπέρ κατά απορρίπτονται 237 υπέρ κατά απορρίπτονται 238 υπέρ κατά αμφίβολο το αποτέλεσμα 238 ηλεκτρονικά ψηφίζουμε 238 Παρακαλώ ψηφίσατε. Υπάρχει κάποιος ε, που έχει χαλαρώσει πολύ. Έχει αποκοιμηθεί. Λοιπόν, από τα 31 ψήφι υπέρ, 39 κατά, απορρίπτεται. Ποιος ξέρει αυτός που κοιμάται πώς ψηφίζει. Λοιπόν, τροπολογία 40. Έχουμε πολύ μακρά τροπολογία υπέρ, κατά, χες, ε, απορρίπτεται. 239 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Όχι. 239. Ε, Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε 239 λοιπόν. ...32 ψήφοι κατά, 38 υπέρ, έχετε δίκιο, αλλά εάν δεν συμμετέχετε, δεν σηκώνει το χέρι, δεν μπορώ να δω. Λοιπόν, 240, εντάφ. υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται, 241. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 242. τίθεται να ελέγξουμε το αποτέλεσμα για το 241. Εντάξει. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για το 241. Δύο κοιμόνται αυτή τη φορά. Κλείνουμε την ψηφοφορία. 32 ψήφοι κατά, 37 υπέρ. Εγκρίνεται. 242 ψήφι Κατά. Απορρίπτεται. 243. Για να κουδάκεις. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Το εκτιμώντας α. 2 ε, και 3 είναι ταυτόσιμες. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Παλέτη. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η 5 έχει αποσυρθεί. Ψηφίζουμε την τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 7. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Υπέρ κατά απορρίπτεται 9 υπέρ κατά <clears throat> απορρίπτεται τροπολογία 10 και 11 είναι ταυτόσιμες τις ψηφίζουμε ομού υπέρ κατά απορρίπτεται τροπολογία 12, 13, 14 είναι ταυτόσιμες ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Απορρίπτονται. 16 υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 15 υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 17 υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 18 υπέρ. Κατά απορρίπτεται 19 υπέρ κατά απορρίπτεται 20 υπέρ κατά απορρίπτεται 21 κοπά υπέρ κατά απορρίπτεται 22 υπέρ κατά απορρίπτεται 23 υπέρ κατά Απορρίπτεται. 24 Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 26. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 26. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 27. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Ψηφιπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Και τώρα η τελική ψηφοφορία επί του τροποποιηθέντος ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία επί του συνόλου του ψηφίσματος, όπως τροποποιήθηκε με την έγκριση των τροπολογιών. Ε, Απίστευτο. Και στην τελική τροπολογία, ε, ψηφοφορία συγγνώμη, υπάρχει κάποιος ε, ο οποίος έχει αποκοιμηθεί. Λοιπόν, 60 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφο κατά. Ομοφωνία. Συγχαρητήρια κυρία εισηγητρία. Έξω από την αίθουσα υπάρχει μια άμαξα με τέσσερα άλογα για να κάνει το γύρο του θριάμβου η κυρία Ρόιτεν. Λοιπόν, περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα που αφορά την έκθεση προόδου της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Εισηγητής ο κύριος Ζόραν Τάλερ. Έχει ζητήσει όμως τον λόγο ο κύριος Τάλερ. Παρακαλώ κύριε Τάλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο των όπως είπα και χτες, και η προσέγγιση στο μακεδονικό ζήτημα έχει συμφωνηθεί μεταξύ των ενδιαφερομένων. Ε, υπήρξαν κάποιες αλλαγές, κάποια αιτήματα μάλλον της τελευταίας στιγμής για ε, διαφορετική διατύπωση. Θα δείτε ότι έχουμε την, πρόταση, έχουμε την πρόθεση μάλλον να διατηρήσουμε το αρχικό κείμενο και εκεί σημειώνουμε το θετικό μας πρόσημο Περιμένω λοιπόν να διεξαχθεί η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Ωραία, με αυτή τη διευκρίνηση μπορούμε να περάσουμε στις ψηφοφορίε. Τροπολογία 1, Γιαννάκο κουμουτσάκο ψηφιπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 2, Χουντή. υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 3, υπέρ, κατά εγκρίνεται 5 η 3 έχει εγκριθεί άρα καταπίπτει η 5, 6 και 7 περνάμε στην 8 ψήφι περ κατά δεκτή 9 υπέρ κατά δεκτή Μπαζέσκου 10 πέρ κατά Απορρίπτεται. Γιαννάκου Μουτσάκος τροπολογία 11. Ψηφιπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Χατζημαρκάκης. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. 13. Γιαννάκου Κουμουτσάκος. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 14. Τροπολογία. Ψηφίζουμε με την προφορική τροπολογία. Ψήφι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. <clears throat> Δεκτή. Συμβαστική τροπολογία 1 του εισηγητή. Ψήφι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Περνάμε στην προφορική τροπολογία 1. Οι υπόλοιπε καταπίπτουν λόγω του ότι ψηφίστηκε η συμβαστική τροπολογία. Ψήφι υπέρ στην παράγραφο 7 της προφορικής τροπολογίας 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ζήτησε τον λόγο η προσυπογράφηση τροπολογία κυρία Κορνέλισεν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να υποβάλω μια προφορική τροπολογία την τελευταία στιγμή για να λάβουμε υπόψη όλες τις ευαισθησίες. Εδώ λέγεται, γίνεται λόγος για μακεδονικές αρχές και παρότι πρόκειται για επίθετο και θα ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθεί αυτός ο όρος, θα θέλαμε να αλλάξει παρακαλώ και να πούμε οι αρχές των Σκοπίων αν δεν έχουν αντίρρηση οι συνάδελφοι συμβαστικά, οι αρχές των Σκοπίων. Ακούσατε την προφορική τροπολογία. Εάν ε, υπάρχουν αντίθετε συνάδελφοι στην τροπολογία θα πρέπει να εγερθούν. Τουλάχιστον έτσι γίνεται στην Ολομέλεια. Όσοι είναι κατά της προφορικής τροπολογίας ας εγερθεί παρακαλώ. Αν υπάρχει σημαντικός αριθμός ε, συναδέλφων που αντιτίθενται τότε δεν θα τη δεχτούμε. Ε, λυπάμαι κυρία Κορδέλης, αλλά δεν μπορούμε να την ψηφίσουμε. Θα ψηφίσουμε την 19 ως έχει στο κείμενο. Δηλαδή με τον όρο μακεδονικές. Ψήφι υπέρ της 19. Κατά. Δεκτή. Τροπολογία 20 Τρεμόπουλος. Εγκρίζει 19, άρα καταπίπτει. Περνάμε στην 21. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία του εισηγητή στην παράφο 8. Προφορική τροπολογία 2. Ψήφι υπέρ. Κατά. <clears throat> Δεκτή. 22. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 23. Περ. Κατά. Δεκτή. 24. Ψήφι υπέρ. Κατά. Νομίζω πως μάλλον εγκρίθηκε. Έχω κάποιες εμβολίες Κουραστήκατε. Κάντε κάποιες ασκήσεις και να σηκώνετε τα χέρια. Προφορική τροπολογία 3 καταπίπτει διότι νεκρή τροπολογία 24. 25 Γιαννάκου Κουμουτσάκος. Μόνο σε ό,τι αφορά τον όρο που αναφέρεται το στο κείμενο urges υπέρ κατά απορρίπτεται. Ας επαληθεύσουμε, εντάξει, ε, τι να κάνω εγώ με δεν ψηφίζετε. Λοιπόν, τροπολογία 25, άρχεται η ψηφοφορία. Μόνο τον, τον όρο ε, urges. Άρχεται η ψηφοφορία. Πάντα έχουμε τον κοιμισμένο. Λοιπόν, 29 κατά 37 υπέρ εγκρίθηκε. Η βασική τροπολογία 2 του εισηγητή υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι τροπολογίες μέχρι την προφορική τροπολογία 4 του εισηγητή. Ψήφι υπέρ της 4. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 31. Υπέρ. <clears throat> Κατά. Εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά δεκτή 34 υπέρ κατά Ας ελέγξουμε καλύτερα. 34. Ψηφίζουμε. Έληξε ψηφοφορία. 38 ψήφοι κατά, 27 υπέρ. Απορρίπτεται. 35. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Συμβαστική 4. Του υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Καταπίπτουν 36, 37, 38, 39 και περνάμε στη 42 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 44 Σαλαβράκος υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 44. Θα επαληθεύσουμε. Τι να κάνουμε, ε, δεν είδα καλά. 44. Ψηφίζουμε επί τη 44. Ηλεκτρονικά. «48 ψήφοι κατά, 17 υπέρ». Άρα απορρίπτεται. 45 Γιαννάκου Κουμουτσάκος. Υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 48 χουντής υπέρ κατά απορρίπτεται. 47 βανόρδεν υπέρ κατά απορρίπτεται. 49 υπέρ κατά εγκρίνεται. 50 υπέρ Ζητώ συγγνώμη. Να έκανα λάθο. Η 50 δεν πρέπει να ψηφιστεί διότι η 49 έγινε δεκτή. Περνάμε στην 46. Όχι. Ούτε. Περνάμε στην συμβασμό 4. Σε χωριστά μέρη. Πρώτο μέρος. Ψηφιπέρ. Κατά. Δεκτό. Δεύτερο μέρος. Περ. Κατά. Δεκτό. 51 καταπίπτει. Καλύπτεται από τη συμβαστική 4 και φτάνουμε στην 57. Ψήφι υπέρ 57. Κατά. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία υπερθμών 5. Νικολάη ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 58. Σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική Πέντε. σε τρία μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Και έτσι καταπίπτει η τροπολογία 59, 60, Μισό λεπτό να διαβουλευτώ με τον γραμματέα. Allora, come indicato nel... αναφέρεται και στον κατάλογο των ψηφοφοριών, η 60 θα πρέπει να ψηφιστεί μέχρι το σημείο όπου αναφέρεται στα σχολικά κείμενα. Ψηφίζουμε την 60. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 61. Τι θέλετε, έλεγχο επί τη 60. Ωραία, εντάξει. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά επί τη 60. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. 24 ψήφοι κατά, 41 ψήφοι υπέρ. Εγκρίθηκε. 61. Όχι. 62. Πλάμψη στην 62. Κατά, υπέρ κατά εγκρίνεται. 32, όχι, όχι, καταπίπτει 32. 63, Σαλαβράκος, υπέρ. Δύο τμήματα πρέπει να ψηφίσουμε. Το πρώτο, ψήφι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Το υπόλοιπο καταπίπτει διότι καλύπτεται από την τροπολογία 60. Λοιπόν, περνάμε στην 64. Δεν ε, ψηφίζουμε 64, 65, 66 διότι καλύπτονται από το συμβαστική 5. Περνάμε στην 67 τελικά. Σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά εγκρίνεται. 68. Όχι, δεν ψηφίζουμε την 68, περνάμε στην 69. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 70. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 71. Υπέρ. Κατά. 72 42 υπέρ, 72 χουντή ε, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 73 Γιαννάκο Κουμουτσάκος υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 74 Σαλαβράκος ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 75. Κοπά, Περ, κατά, απορρίπτεται. 76, να κουκουμουτσάκο, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 78, 77, συγγνώμη, χουντή, υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτεται. 78, δεν τη ψηφίζουμε διότι είναι ταυτός με 77, 79, Γιαννάκο Κουμουτσάκος, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 80, κατά εγκρίνεται 81 υπέρ κατά εγκρίνεται 82 κοπά υπέρ κατά δεκτή λοιπόν θα ψηφίσουμε τώρα την τροποποιητής ε, πρόταση στο σύνολό τη άρχιτη ψηφοφορία Si chiude la votazione. 56... Πέρα ψηφοφορία, 56 ψήφοι υπέρ, 5 ψήφοι κατά, συγχαρητήρια στον εισηγητή, α και 5 αποχές. 5 κατά και 5 αποχές. Εγκρίνεται. Λοιπόν, η πρόταση ψηφίσματος και τώρα περνάμε στην ψηφοφορίες αναφορικά με την πρόοδο της Κροατίας το 2009. εισηγητής είναι ο κ. Βόμπολα. Παράγραφος 1, τροπολογία 12, 4 μέρη. Ψήφι υπέρ του πρώτου μέρους. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία του εισηγητή ψήφι υπέρ. Υπέρ κατά. Απορρίπτεται. Ε, δεκτή τέταρτο τμήμα υπέρ κατά Φαίνεται πως εγκρίνεται, αλλά παρακαλώ να συμμετέχετε. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 15 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος πρώτη υπέρ κατά δεκτό. Δεύτερο μέρος. Α, θέλετε πάλι δύση, ωραία. Πρώτο μέρος τροπολογίας 15. Άρχεται η ψηφοφορία. 18 κατά 40 υπέρ. Δεν ψηφίζεται. Περνάμε στο δεύτερο μέρο, Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ναι. Ψηφίζουμε για το δεύτερο τμήμα ηλεκτρονικά. Τροπολογία 15 δεύτερο τμήμα. Ηλεκτρονικός Λοιπόν, 32 κατά, 29 υπέρ, απορρίπτεται. Προπολογή 16 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 17 υπέρ, κατά, δεκτή. 19 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 18 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 20 υπέρ, κατά, Αγκρίνεται. 21 υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβαστική ένα του Πρώτο τμήμα υπέρ. Ο Σβόμπολα θέλει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα το δεύτερο τμήμα να το αποσύρω. Για τον εξή λόγο. Χτε ε, το συζητήσαμε. Αυτό που λέμε για την πλήρη συνεργασία με το ΕΙΚΤ αναφέρεται και στο πρώτο τμήμα και στο δεύτερο τμήμα μας ανέφερε ο κ. Μπρέμετ ότι δεν ξέρει καν και ο ίδιος αν υπάρχουν τα έγγραφτα. Γι' αυτό λοιπόν να αποσύρουμε το δεύτερο τμήμα. Να... Γιατί αν αναφέρεται η αναφορά για, την, για, τα, για τη συνεργασία, την πλήρη συνεργασία και στο πρώτο τμήμα. Εντάξει. Ψηφίζουμε το πρώτο, το τρίτο και το τέταρτο. Πρώτο το υπέρ, κατά δεν κρίνεται. Δεύτερο δεν ψηφίζουμε. Το τρίτο υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Λοιπόν, αυτή η συμβασική τροπολογία οδηγεί στο να καταπέσουν ε, αρκετές τροπολογίες και φτάνουμε στην 26. Ψήφι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά, απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία του εισηγητή. Ψήφ υπέρ. Κατά ε, εγκρίνεται. Τροπολογία 29, 28 καταπίπτει. ψήφ υπέρ της 29. Κατά απορρίπτεται. 31. Πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Νομίζω πως εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 30. Υπέρ. Κατά. Ασαφές το αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε την 30 ηλεκτρονικός. Μας λείπουν δύο ψήφοι. Και, και η γνωστή, ο γνωστός υπόπτος. Λοιπόν, 30 ψήφοι κατά, 29 υπέρ. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 32. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. 34 καταπίπτει. Πρέπει να ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία 3. Ψήφι υπέρ της προφορικής 3. Κατά. Δεκτή. 35 καταπίπτει. Περνάμε στα συμβαστική 2. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 36 σε τρία τμήματα, αλλά εγκρίθηκε συμβαστική 2, οπότε καταπίπτει. Περνάμε στην 37. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. 38. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. 39. Υπέρ κατά απορρίπτεται 40 σε δύο μέρη πρώτο μέρος υπέρ κατά απορρίπτεται δεύτερο μέρος υπέρ κατά απορρίπτεται 41 υπέρ κατά απορρίπτεται 42 υπέρ κατά απορρίπτεται 43 υπέρ κατά εγκρίνεται παράγραφος 45 συγγνώμη 25 τροπολογία 44 πρώτο μέρος υπέρ κατά απορρίπτεται δεύτερο μέρος υπέρ κατά απορρίπτεται 45 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 47 υπέρ. Κατά. Νομίζω πως εγκρίθηκε. 48 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ. Το πρόβλημα έχει αποσυρθεί, Πρόεδρε. Με έχει αποσυρθεί από τους πράσινους. Α, ναι, ναι, έχετε δίκιο. Το γράφει και εδώ. Withdrawn by the Greens. Συγγνώμη, δεν το διάβασα. Μου διέφυγε. Δεύτερο μέρος, λοιπόν, τη 48 υπέρ. Κατά ασαφές το αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα της 48. Άντε άλλος ένας. Λοιπόν, 25 ψήφοι κατά, 31 ψήφοι υπέρ, εγκρίνεται. 49 ψήφοι υπέρ κατά δεκτή 50 υπέρ κατά εγκρίνεται και τώρα πάμε στα εκτιμώντας τροπολογία 2 υπέρ κατά υπορρίπτεται 3 υπέρ κατά δεκτή 4 υπέρ κατά απορρίπτεται 5 υπέρ κατά απορρίπτεται 6 υπέρ κατά απορρίπτεται 7 υπέρ κατά απορρίπτεται συμβιβασμός 3 του εισηγητή υπέρ κατά δεκτός ε, καταπίπτουν οι τροπολογίες ε, που ακολουθούν μέχρι την 11 που ψηφίζουμε σε τρία μέρη. Πρώτο μέρος ε, ψηφιπέρ. Κατά απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά απορρίπτεται. Τρίτο μέρος υπέρ κατά απορρίπτεται. Το τροπολογία 1 του λοιπόν, υπέρ κατά δεκτή και η τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροποποιηθήσα έκθεση. να σας ανακοινώσω με ιδιαίτερη χαρά πως ο, ο μας που είχε αποκοιμηθεί ξύπνησε 62 παρόντες, 62 ψηφίσαντες. Καλά στα ξυπνητούρια. 54 λοιπόν υπέρ, καμία ψήφος κατά, 8 αποχές. Σε χαρακτήρια στον εισηγητή. Και περνάμε στην τελευταία για σήμερα ψηφοφορία που αφορά στην έκθεση Σάιρους Βόλσκι για την ασφάλεια του εφοδιασμού σε φυσικό αέριο. Περνάμε στον συμβασμό υπαρθμών 1, ψηφιπέρ, κατά, δεκτός. Περνάμε στην τροπολογία 38 υπέρ, κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά δεκτή. Τροπολογία 40 υπέρ κατά δυστυχώς απορρίφθηκε. Τροπολογία 40 ε, 7 συγγνώμη σε τρία μέρη. Πρώτο μέρος, υπέρ. Κατά. Δεκτό. Δεύτερο μέρος, υπέρ. Κατά. Δεκτό. Τρίτο μέρος, υπέρ. Κατά. Δεκτό. Συμβασμός 2 του εισηγητή υπέρ. Ψήφι κατά. Εγκρίνεται. Έτσι καταπίπτουν οι τροπολογίες που ακολουθούν έως τον συμβαστική 3 ψήφι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Περνάμε στον συμβιβασμό 4, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Περνάμε στην 45, Χατζηγεωργίου, υπέρ, κατά, Α, απορρίπτεται. 10, υπέρ, κατά, δεκτή συμβαστική 5 του εισηγητή ψήφι υπέρ κατά από εγκρίνεται. 47 τροπολογία υπέρ κατά εγκρίθηκε. Χαίρομαι. 12 υπέρ κατά εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά εγκρίνεται. 48 Χατζηγεωργίου υπέρ κατά απορρίπτεται 17 υπέρ κατά δεν εγκρίνεται 16 υπέρ κατά δεκτή 49 υπέρ κατά εγκρίνεται 17 υπέρ κατά εγκρίνεται 50 Χατζηγεωργίου υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αγκρίνεται. Έτσι καταπίπτουν οι τροπολογίε 51 και 18. Περνάμε στην 52 υπέρ. Κατά. Ε, ναρκισιστικά το βάζω, το θέτω σε ψηφοφορία. Δεν είναι, δεν σηκώσατε το χέρι. 52. Λοιπόν, ψηφίζουμε την 52 ηλεκτρονικά άρχη ψηφοφορία. Να, θα ιτηθώ, θα ιτηθώ. Δεν σηκώσατε τα χέρια σας για λόγους ευγένεια. Έληξε η ψηφοφορία 52. Ε, πω, με διαλύσατε. 35 ψήφικα κατά, 19 υπέρ. Με ταπεινώσατε. Ε, κατά τα άλλα υπαθέστατη. 53 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 54. Είναι, συ... είναι συμβατή με 53. Δεν αναφέρεται καν κάποιο πρόσημο θετικό ερευνητικό. Λοιπόν, 54 ψήφι υπέρ. Υπέρ. Άντε, άντε. Κάντε κάτι. Ψήφι κατά. 19 του εισηγητή. Υπέρ. εγώ Εγωιτήθηκα φυσικά. Ε, 50, εγκρίθηκε. 55 καταπίπτει. 56 Χατζηγοργίου υπέρ. Κατά να απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 57 Χατζηγοργίου Χουντής υπέρ. Κατά απορρίπτεται. Ε, η 58 έχει αποσυρθεί. Ψήφι υπέρ της του συμβασμού μετά. δεν γίνεται δεκτός και έτσι καταπίπτουν μια σειρά από τροπολογίες, φτάνουμε στην 63. Όχι, γιατί στην υπέρ, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ο, 23 υπέρ κατά 24 Χατζηγεωργίου υπέρ κατά απορρίπτεται 25 Χατζηγεωργίου χουντίσο υπέρ κατά εγκρίνεται 8 συμβασμός του εισηγητή υπέρ κατά δεκτή δεκτός Περνάμε στο συμβασμό υπαρχμών 9, τα προηγούμενες δύο έχουν καταπέσει, ψήφι υπέρ, κατά, Δεκτός, περνάμε στην τροπολογία 28, Χατζηγεωργίου Χουντής, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβασμός 10, υπέρ, κατά, Αγκρίνεται. Φτάνουμε στο συμβασμό 11, σε δύο μέρη, πρώτο μέρος, υπέρ, κατά, δεκτό, δεύτερο μέρος, υπέρ, κατά, δεκτό. Τροπολογία 30, 31 και 4 Περνάμε στην 33. Τα παραπάνω καταπίπτουν. 33. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Λαντσμπέργες 34 καλύπτεται από το Σύμβασμο 11 και η 35 επίση ε, χωριστή ψηφοφορία συνολική ψηφοφορία, συγγνώμη, ε, το, επί της τροποποιηθής σας ε, έκθεσης, ε, άρχεται ψηφοφορία. Τρεις συνάδελφοι απουσιάζουν από την κλίση. Μάλλον άφησαν το... την κάρτα του στο μηχάνημα αφού αναχώρησαν από την αίθουσα. Εμπεστώσει έχουμε 47 ψήφους υπέρ, 4 ψήφους κατά και μία η αποχή. Συγχαρητήρια κύριε Ισηγητά. Η ασφάλεια του εφοδιασμού σε φυσικό αέριο έγινε δεκτή να υπογραμμίσω συγχαίροντας τους συναδέλφους ότι ολοκλώσαν οι ψηφοφορίες ακριβώς στις 10 και 30. Νομίζω πως η ΝΑΣΑ κυβερνά και διευθύνει αυτή την αίθουσα. Bene, qualche minuto Να δώσουμε λίγο χρόνο στους συναδέλφους ε, και τους υπολείπους που επιθυμούν να εγκαταλείψουν την αίθουσα προκειμένου να το πράξουν ησύχως ε, και μπορούμε να περάσουμε στη συζήτηση για το θέμα της απαλλαγής 2008, γενικός απολογισμός ε, Τμήμα 3, Επιτροπή. Η ε, και συντάκτης είναι ο κύριος Γκάλερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να μην περιμένουμε λίγο όμως μέχρι να βγει ο πολύς ο κόσμος και να έχει επανέλθει λίγο η ησυχία. Come vuole, possiamo aspettare qualche minuto, non siamo in ritardo. Siamo stati... Εντάξει, επειδή ήμασταν πολύ ακριβείς μέχρι τώρα, μερικά δευτερόλεπτα μπορούμε να περιμένουμε. Παρακαλώ συνάδελφοι που ετοιμάζετε να εγκαταλείψετε την αίθουσα, φροντίστε να το πράξετε. Δεν χρειάζεται να συζητάτε εδώ τις προσωπικές και ιδιωτικές συζητήσεις. Μπορείτε να το πράξετε έξω από την αίθουσα και να είστε κι εσείς καλά και εμείς καλύτερα. Κύριε Γκάλερ, νομίζω ότι έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις για να συνεχίσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλάμε λοιπόν εδώ για την ε, γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτορικών Υποθέσεων για την χορήγηση απαλλαγής για τον προπολογισμό του 2008. Έγιναν πληρωμές σε ύψος περίπου 5 δισεκατομμυρίων ευρώ και το ελεγκτικό συνέδριο διαπιστώνει στα πορίσματά του ότι υπήρχαν κάποιες ανακρίβειες σε ορισμένες περιπτώσεις και ότι τα συστήματα εποπτείας και παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξωτερική βοήθεια, την αναπτυξιακή βοήθεια, ε, εν μέρη ε, απέβησαν μία αποτελεσματικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποδεικνύει τον ιδιαίτερο τρόπο εργασίας του ελεγκτικού συνεδρίου που βλέπει με την αιτήσια παρακολούθηση μόνο ένα κομμάτι της εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε ό,τι αφορά όμως ε, τα περισσότερα ε, ευρωπαϊκά προγράμματα διαμορφώνονται σε βάθος χρόνων και υπάρχουν διορθωτικοί μηχανισμοί οι οποίοι όμως επιτρούν επί όλου του κύκλου και όλες τις διάρκεια των προγραμμάτων. Το ελεγκτικό συνέδριο πρέπει ωστόσο να διεξάγει αξιόπιστη και ανεξάρτητη έρευνα. Ωστόσο, το ελεγκτικό συνέδριο κρίνει αρνητικά σε ό,τι αφορά την εξωτερική βοήθεια, την απτυξική βοήθεια και την ε, διεύρυνση, αλλά συνολικά το περιθώριο εσφάλματος, επειδή έγιναν ε, ε, βελτιώσεις και διορθώσεις, είναι περιορισμένο. Και το ελεγκτικό συνέδριο σε ό,τι αφορά την κανονικότητα και την ε, ορθότητα της μεθοδολογίας, μεθοδολογίας διαπιστώνει ένα περιθώριο 2-5% της δειγματοληψίας. Τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα από ότι στην πολιτική συνοχής. Αν θα το παρακαλώ να κάνατε ησυχία. Αυτό το περιθώριο σφάλματο λοιπόν 2 5% δειγματοληψία διαπιστώνεται στον δικό μα τομέα. Καλύτερα τα πράγματα από ότι στον τομέα τη πολιτική συνοχή και παρόμοια τα πράγματα όπω στον ε, ε, κλάδο τη έρευνα, τη ε, μεταφορά και το καθεξή. Και προφανώ ε, παραμένουν κάποια προβλήματα σε ό,τι αφορά τους ελέγχους. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τους ελέγχους και τις παρατηρήσεις που έγιναν από το ελεκτικό συνέδριο θα πρέπει να τις λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε ό,τι αφορά τις συστάσεις του ελεκτικού συνεδρίου. Στην πρότασή μου για την γνωμοδότηση της ε, Επιτροπής μας αναφέρω τα βασικά έξοδα τα βασικά μέσα σε ό,τι αφορά τον δικό μας πολιτικό κλάδο και είμαι πρόθυμος να συμπεριλάβω περαιτέρω σχόλια των συναδέλφων, αλλά σε ό,τι αφορά τους χαρακτήρες της ε, γνωμοδότησής μου είμαι κάπως περιορισμένος, δεν έχω α, απεριόριστα απεριόριστο χώρο, αλλά θα τις κοιτάξω τις ε, εισηγήσει των συναδέλφων. Κατέκτησα το κείμενο στα αγγλικά, τα συνόψισα σε πέντε τμήματα. Στον πρώτο τμήμα αναφέρω ότι καλώς ορίζει τι αντικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια του στόχου και τη ε, διεθνή συντονισμό των δονητών που επέφερε η ίδρυση του μηχανισμού Πήγασος που αναπτύχθηκε σε βάση με τη βάση του εργαλείου TIM. Ξέρετε ότι πρόκειται για ένα νέο μέσο χρηματοδότηση τη Παλαιστινιακή Αρχή. Στο δεύτερο, ότι σημειώνει την τάση αυξανόμενων ε, συμβολών σε ταμεία πολλαπλών δωρητών και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον ΟΗΕ, ωστόσο αναφέρει την ε, ε, έλλειψη ικανοποίηση σε ό,τι αφορά τα συνεχιζόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ελεγκτικό συνέδριο σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα χρηματοοικονομικά κείμενα, ε, έγγραφα των ε, υπηρεσιών του ΟΗΕ και στο επόμενο σημείο αναφέρεται ότι σημειώνουμε τη συστάσεις του δικαστηρίου σε ό,τι αφορά τους στρατηγικούς στόχους και το καθεξής. Μετά έχουμε την ειδική έκθεση παριθμών 16 του 2009 για την Τουρκία, όπου καλύπτεται η περίοδος πριν την εφαρμογή του μέσου για τα προενταξιακή βοήθεια και αναφέρονται οι θετικές εξελίξεις που επέφερε το μέσο αυτό, ωστόσο τονίζεται πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη και ορθή εφαρμογή του μέσου ΕΠΑ, IPA. Και όλα αυτά θα πρέπει φυσικά να ληφθούν υπόψη. Τελευταίο στοιχείο, σημείο, σε ό,τι αφορά την ε, χρηματοδοτική υποστήριξη πέρα από άλλα μέσα για την ενίσχυση της ιδιοκτησίας στην χώρα, αλλά φυσικά θα πρέπει να συνοδεύεται το μέσο αυτό από σαφείς στρατηγικές και σαφείς μηχανισμούς ελέγχου προκειμένου να επιλεφθούν οι συγκεκριμένες απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τις πληρωμές και τους συγκεκριμένου όρους αναφορικά με τους αποδέκτες της βοήθειας. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αποστείλουμε ως γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Μπορούμε να περάσουμε στη συζήτηση. Ο κύριος Μπρόκ έχει λόγο. Πρόεδρε. Παρακολούθησα με πολύ ενδιαφέρον και ικανοποίηση την έκθεση του συναδελφού Γκάλλαρ. Αν και βλέπω ότι δεν έχουμε τόση έμφαση δώσει προς την ε, πολιτική της συνοχής ως προς εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της κυρίας Φρέρο Βάλτερ της ε, προηγούμενης ε, Επιτρόπου. αυτή. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα πολύ ευρύτερο ότι δεν ε, έχουμε αξιοποιήσει την πολύ σοβαρή ε, δυνατότητα ελέγχου μας προσφέρει από το 1999 το νέο σύστημα έστερα από την αποτυχία της Επιτροπής ε, Σαντέρ και εδώ βλέπουμε σε πολλούς τομείς και εδώ αλλά και σε άλλους τομείς πολιτικής ότι το σύστημα αυτό είναι πολύ βαρύ και ίσω με τη νέα επιτροπή που περιμένουμε τώρα να λάβει καθήκοντα θα μπορούσε και ο κύριο Γκάλερ να εξετάσει και τι πτυχέ των εξωτερικών ε, σχέσεων βεβαίω, αλλά και το δημοσιονομικό πλαίσιο. Ξέρω και ότι και οι συνέδελφοι από τον, ε, την Επιτροπή Ελέγχου του ίσω να μην είναι πολύ ε, ευτυχεί στο να ακούνε πράγματα, αλλά πολλέ φορέ έχει τεράστια σημασία ο παράγων χρόνο σε αυτές τις υποθέσεις εξωτερικές σχέσεις. Μπορεί να αλλάξουν πολλά εάν καθυστερήσουμε λίγο και το είναι τόσο βαρύ το σύστημα. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι η Επιτροπή ήδη έχει προχωρήσει τόσο που υπάρχει και, έχει και προσωπική ευθύνη ένας Επίτροπος, ε, εμείς το να μην έχουμε ικανοποιητική, το να διαπιστώνουμε ότι δεν είναι επαρκής η αποτελεσματικότητα των δράσεών μας, είναι πολύ ανησυχητικό. Και ναι, μεν θα υποστηρίξω την απαλλαγή, όπω ο Κύριο Γκάλερ, αλλά θα πρότεινα να γίνει μια έρευνα για το πώς θα μπορούσαμε καλύτερα στο μέλλον να ε, ε δρούμε στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων. Και θα ήθελα να το συστήσω αυτό και με του αδέρφου της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού. Ευχαριστώ κύριο Γκουαλκέρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω πως συμφωνούμε απολύτως με τις κατευθύνσεις γραμμές της έκθεσης Γκάλερ, με την ανάλυση που κάνει και με τις βελτιώσεις που προτείνει για κάποιους μηχανισμούς χρηματοδοτικούς των σχεδίων, την αξιολόγηση κάποιων προγραμμάτων κάποιων προβλημάτων που υφίστανται και τη δυνατότητα να μπορέσουν να ξεπεράσει το θέμα της ΦΑΦΑ. Ευχαριστώ. Αυτά. Η κυρία Μπράτν έχει το λόγο. Ευχαριστώ και σε ευχαριστώ επίση ε, για τον κύριο, προς τον κύριο Γκάλερ για την έκθεσή του. Και θέλω όπω και ο κύριος Μπροκ να δω και θα καταθέσουμε και τη σχετική τροπολογία, αλλά δεν ξέρω ως εισηγήτρια για το ε, μέσο σταθερότητας βλέπω ότι πολλά είναι τα ε, μέσα ή τα προγράμματα τα οποία προχωρούν θα μπορούσαν να έχουν χρηματοδοτηθεί από άλλα μέσα, πριν όμως χρηματοδοτούνται από το μέσο σταθερότητα γιατί είναι πιο ευέλικτο αφενός και αφετέρου πράγματι υπάρχει δυνατότητα τα χρήματα που δεν να τα αξιοποιήσουν οι παράγοντες επιτόπου στην ουσία. Γι' αυτό λοιπόν σημειώνω ότι υπάρχουν ζητήματα ως προς την εφαρμογή, ως προς την χρήση των ε, κονδυλίων. Και θα ήθελα να ε, εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ευελιξία ως προς ε, τμήματα τουλάχιστον των μέσων, των χρηματοδότηση που διαθέτουμε, μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να παρεμβαίνουμε πιο αποτελεσματικά, ώστε να μην φτάνουν τα χρήματα εκεί που θέλουμε να τα διαθέσουμε όταν πια είναι πάρα πολύ αργά. Τώρα παρακαλώ τον λόγο να λάβει ο Δόκτωρ Μίλερ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε λεπτομερή σχόλια να κάνουμε ως προς την έκθεση του κυρίου Γκάλερ, την ομοδότησή του. Ευχαριστούμε για τις επικοδομητικές προτάσεις που ετυπώνει. Μπορούμε να κάνουμε δεκτές την πλειονότητα τους, της ε, προτάσεις του κυρίου Γκάλερ. Τις περισσότερες μάλιστα ήδη τις έχουμε θέσει εφαρμογή και η κυρία Φεροβάλτνερ είχε ήδη φροντίσει και να, να έρθει σε επαφή με τον κύριο Γκάλερ και είναι βέβαια στη θέση της Επιτροπής ε, για να απαντήσει οποιασδήποτε ερωτήσει. Ευχαριστώ. Σαλαφράγκα. Ο κύριο Σαλαφράγκα ζήτησε καθυστερημένα τον ε, λόγο, αλλά πάση παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε, δεν νόμιμη, δεν ξέρω ότι θα βιαζόσατε να δώσετε το λόγο στην ε, Εκπαιδευτική Επιτροπή. Ε, νομίζω πως η έκθεση του κυρίου Γκάλερ είναι πολύ καλή, είναι ε, κάπως επικριτική αλλά επικοδομητική και θέτει το θέμα στην πολύ σωστή διάσταση. Συχνά το ζήτημα της απαλλαγής χρησιμοποιήθηκε από πολιτικής ε, πλευράς ενάντια στην Κομισιόν. Η κυρία Βάλτνερ ε, θεωρώ ότι έκανε μια δουλειά πάρα πολύ καλή και κατέδειξε τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να δαπανώνται σωστά τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εξωτερική πολιτική. Ο κ. Μπρόκ έθεσε ένα ζήτημα που ξεπερνάει αυτό το ζήτημα του απαραγής του 2008 και μίλησε για την αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και νομίζω η Πρόεδρε πως ε, κάποια στιγμή θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό, να προβληματιστούμε στην Επιτροπή μας σχετικά με την αποτελεσματικότητα αυτής της ε, βοήθειας μετά από την κατάρρευση της ε, Επιτροπής υπό τον Σαντέρ ξέρουμε ότι σιγά σιγά τα πράγματα άλλαξαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ανακαταστήκαμε πολύ πιο αποτελεσματικοί στην εξωτερική βοήθεια. Με πάση περιπτώσει αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα το οποίο ξεπερνάει κατά πολύ το ζήτημα της απαλλαγής ε, για το 2008 και θα ήθελα να παραμείνω σε ένα σημείο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό το τονίζει ο κύριος Γκάλε στην έκθεσή του, η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν συνεισφέρει με τεράστια ποσά στα διάφορα ταμεία του ΟΗΕ. Εγώ δεν έχω τα ποσά μπροστά μου, αλλά πρέπει να είναι της τάξης του 1300, μάλλον 1 δις 300, 1 400 δισεκατομμύρια ετησίως. Θα πρέπει λοιπόν ε, αυτό να το έχουμε υπόψη μας και θα πρέπει να φροντίσουμε να ελέγχουμε την ε, χρηστή χρησιμοποίηση αυτών των ποσών. Η έκθεση λοιπόν του κ. Γκάλερ είναι πολύ σωστή και θα πρέπει να καταδείξουμε μεγάλη ευαισθησία πάνω στο θέμα, διότι ποσότητες χρημάτων τόσο σημαντικές να γνωρίζουμε πού πηγαίνουν και αυτό όχι μόνο εμείς αλλά να το γνωρίζει και ο Ευρωπαίος Φορολογούμενος. Ευχαριστώ κύριε Σαλαφράγκα. Το λόγο για τα τελικά σχόλια έχει ο συγητής Γκάλερ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους. η συζήτηση αυτή για την ε, απορρόφηση των κονδυλίων, ταχεία απορρόφηση των κονδυλίων, έχει γίνει πολλές φορές εδώ στην Επιτροπή μας εδώ και πολύ καιρό και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει η εξωτερική πολιτική, επί παραδείγματι, να μην συγκρίνεται με, μια, με τη γεωργική πολιτική. Έχουμε Ε, για τη γεωργική πολιτική σε θέσή μας ακόμη και τους δορυφόρους για να βλέπουμε εάν είναι τα αγροτεμάχια εξίσου μεγάλα και η παραγωγή της ε, ελιάς του σίτου εκτεταμένη στην επιφάνεια την οποία ισχυρίζεται ο γεωργός. Αυτά όμως ε, τα μέσα δεν τα έχουμε στη θέση μας για την εξωτερική πολιτική όταν αναλαμβάνουμε είτε στο Ιράκ είτε στο Σουδάν είτε σε άλλους τομείς, σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ανάγκη για κατεπίγουσα βοήθεια Πρέπει να είμαστε σε θέση να διαθέσουμε αμέσως τα κονδύλια εκεί που χρειάζονται. Και πρέπει νομίζω να δούμε πόσο ε, θα εξασφαλίσουμε περισσότερη ευελιξία για τα κονδύλια αυτά. Όπως είπα και για τον κύριο Σαλαφράγκα, θα συμφωνήσω μαζί του. Θα πρέπει αυτό το λεγόμενο ΦΑΦΑ, το Δημοσιονομικό Πλαίσιο Συνεργασίας, ε, να το ε, συμφωνήσουμε με τα Ηνωμένα Έθνη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και φυσικά εννοώ ότι αυτό είναι καθήκον της Επιτροπής, όχι του Κοινοβουλίου. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Να σα πω μερικά θέματα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα. 8 ε, Φεβρουαρίου είναι η καταρχική προβλήμα για την ε, κατάθεση τροπολογίων, 16 Μαρτίου θα εξετάσουμε τα ζήτημα στην Επιτροπή μας και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα περάσει από το Ολομέλεια του Απριλίου. Περνάμε στο επόμενο σημείο της Μεσής Διατάξεως σχετικά με τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για συνεργασία με τις ε, ευβιομηχανισμένες χώρες τροποποίηση του κανονισμού Ευρωπαϊκή κοινότητα 1934 κάθετο 2006. Το λόγο έχει η κυρία Λοκ Μπίλερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στην τελευταία νομοθεσία είχε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Επιτροπή μας ε, να ε, δημιουργήσει ένα νέο όργανο για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες των αναπτυσσομένων χωρών που δεν καλύπτονται από την αναπτυξιακή συνεργασία. Και επίσης είχαμε ζητήσει, είχαμε προτείνει να μετατραπεί το υφιστάμενο μέσο για τις βιομηχανικές χώρες ως σε μέσο συνεργασίας ε, με τρίτες χώρες εκτός των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι θα μπορούσαμε το αναθεωρημένο μέσον αυτό να δράσουμε καλύτερα και να έχουμε και τις σχετικές ε, αλλαγές και στον τίτλο και γι' αυτό αλλάξαμε τον τίτλο αποκολώντας το δημοσιονομικό μέσο για την κάλυψη των αναγκών των, ε, ε, των μη αναπτυξιακών αναγκών των κρατών της Αφρικής, της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής. MAAS θα ήταν τα αρχικά του, άμας δηλαδή. Νομίζω ότι είναι καλύτερο όταν έχουμε το θέμα αυτό προ να είναι και η συντομογραφία του τέτοια που να μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε εύκολα. Ήρθαμε, είδαμε λοιπόν μετά τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Επιτροπή Εξωτερικού Εμπολίου ε, κατουσία, ως κατουσίαν αρμόδια γιατί είναι για λόγους αρικούς εκείνη η οποία έχει αρχικά αναλάβει το πακέτο ICI. Η ΑΦΕΤ ζήτησε να της επιτραπεί η δυνατότητα της να αναλάβει καθήκοντα ε, συνεργαζόμενης επιτροπής ε, γιατί δεν θα είχε μόνο να αναλάβει την προσπάθεια για διορθώσεις στο αρχικό μέσο, αλλά και να χαράξει αρχικές, ε, σε αρχική φάση τις σχέσεις εξωτερικής συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης αφενός και ε, Ασίας, Λατινικής Αμερικής, Αφρικής και Μέση Ανατολής αφετέρου. Προσδιορίζεται λοιπόν το πλαίσιο των αρχικών 17 κρατών υψηλού εισοδήματος του IC e και των λοιπόν 46 που καλύπτονται από τον κανονισμό DCI και προτείνεται να διπλασιαστεί το, ποσοστό, το ποσό αναφοράς για τη συνεργασία που προτείνεται από τα 172 εκατομμύρια στα 148 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2010-2013. Από την θέση ισχύ της συνθήκης Λισαβόνας η, νέα, η νομική βάση ε, χρειάστηκε να τροποποιηθεί για τον αυτόνομο ε, μέσον. Γίναν διάφορες διαβουλεύσεις ως προς την νομική βάση και όπως αναφέρεται και στην πρώτη τροπολογία άλλωστε, προτείνουμε αυτό το οποίο μας έχουν υποδείξει νομικές μας υπηρεσίες. Η πρώτη λοιπόν τροπολογία αναφέρει ότι δεδομένων των όσων προβλέπει η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερο στο άρθρο 212, 207, δεύτερη παράγραφος και 209 παράγραφος 1 κτλ. Στη δε επιτροπολογία τώρα. Το πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, το Μέσο για την Αναπτυξιακή Συνεργασία, όπως και το Μέσο Σταθερότητας, έχει θεωρηθεί από την ΑΦΕΤ και την ΔΕΒΕ ότι θα πρέπει να ε, εξετάζονται ως ε, ως κατεντολήν ε, καθήκοντα των, ε, των εξωτερικών σχέσεων υπό το άρθρο 209. Γι' αυτό θέλαμε την αναδιαμόρφωση του αρχικού μέσου ICI, ε, πράγμα το οποίο θα επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προβάλλει αντιδράσει ω προ τα σχέδια πολιετού συνεργασία, τα προγράμματα πολιετού συνεργασία, εάν το έκρινε απαραίτητο. Τη θέση αυτή υιοθέτησε και η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου, την απέρριψε όμω η νομική υπηρεσία των άλλων διαθεσμικών οργάνων. Και έτσι οι τροπολογίες που έχουμε εδώ στο κείμενό μας που έχουν να κάνουν με την ε, κατεχώρηση κατά πληρεξουσιο, εξουσιοδότηση ΕΚΤΣ θα είναι μόνο αυτά τα οποία μπορούμε να προβάλλουμε. Χαρακτήρας του μέσου αλλάζει από ένα μέσο που ε, υποβοηθά μόνο οικονομικές και εμπορικές σχέσεις, ένα μέσο που βοηθά, που αρχικά ήταν για τις, απευθυνόταν στις πιο εύρωστες οικονομικά χώρες, τώρα προχωράει σε ένα μέσο για την υποστήριξη των αναπτυσσόμενων και φτωχότερων χωρών. Με τη νέα του αυτή μορφή το μέσο θα πρέπει να περιλαμβάνει και κοινωνικά, πολιτικά, ε, οικονομική, κοινωνική και πανεπιστημιακή και συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητών και έχουμε να κάνουμε λίγο πολύ με τις χώρες στόχου που ονομάζονται χώρες εταίροι. Διότι οι βιομηχανικές χώρες, ε, οι πιο εύρωστες οικονομικά, είναι λιγότερες του ενός τρίτου του συνόλου των ε, κρατών ε, δικαιούχων και αυτό θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε στο κείμενο, όπως άλλως θα πρέπει και να γίνει σε διάκριση μεταξύ του DCI που θα πρέπει να χρηματοδοτεί την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, ενώ το νέο μέσων, με την, των βιομηχανικών χωρών, με την αναμόρφωσή του, θα πρέπει να καλύπτει άλλα ζητήματα και πάντως όχι αναπτυξιακά. Στην υπαριθμόν 7 υπογραμμίζουμε το τι θα στοχεύει αυτή η συνεργασία. Ως στόχους λοιπόν ορίζουμε. Το είναι ενίσχυση του διαλόγου με τις χώρες που ε, θα πραγματοποιηθεί με τον ε, διάλογο, την ανταλλαγή, τις ανταλλαγές και τη συνεργασία. Προαγωγή της επιστημονικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας σε διάφορους τομείς. Προαγωγή ε, θεμητών συνθήκων ε, οικονομικής συνεργασίας και συναλλαγών σε πάντα προσαρμοσμένων και στους στόχους χιλιετίας, ενίσχυση των ανταλλαγών με τις ε, χώρες εταίρους, εσωματωσή τους σε πολυμερή κέντρα συζητήσεων, ανάπτυξη των ε, συζητήσεων για την αντιμετώπιση των πολυμερών προκλήσεων όπως κλιματική αλλαγή, ασφάλεια της ενέργειας, ειρήνη και ιδιαίτερη έμφυση στις ε, στις βιώσιμες τεχνολογίες, οι αηφόρε τεχνολογίε, σεβασμό των πνών δικαιωμάτων τη δημοκρατια των θεμελιωδών ελευθεριών, του κρατου δικαίου, τη ε, χρυση διακυβερνηση ισοτιμη ε, και δικαιη οικονομικη και εμπορική αναπτυξη κοινωνικη προστασια και ιδιαίτερη προστασία των μειονοτήτων. Μέχρι στιγμη η αλλαγή του πεδίου εφαρμογής του μέσου είναι αυτή που σας ανέφερα μέχρι τώρα και κλείνοντας θα ήθελα να αφαιρθώ στα οικονομικά στοιχεία. Όπως αναφέρεται εξ αρχής, η Επιτροπή έχει προσθέσει 176 εκατομμύρια ε, ευρώ για τις νέες χώρες, επιπλέον των 172 εκατομμύριων ευρώ που προβλέπονταν αρχικά και θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι τα χρήματα αυτά θα θέλαμε να είναι ε, πιο αναλογικά ως προς τις ανάγκες των κρατών που βλέπουμε εδώ. Γι' αυτό προτείνουμε από τα 448 εκατομμύρια ευρώ τα 2 τρίτα να κατανεμηθούν σε χώρες που έχουν πραγματικά ανάγκη και το 1 τρίτο στις χώρες του παραρτήματος ε, υπαριθμών 1, δηλαδή χώρες ε, με υψηλό εισόδημα. Επίσης θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι θεωρώ ευπρόσδεκτη την τοποθέτησή του εισηγητού της Σύντρα και της ΔΕΒΕ ότι δεν πρέπει να υπάρξει πρόσθετη χρηματοδότηση από το TCI και προτείνουμε στην τροπολογία μας να αναζητηθεί πρόσθετη χρηματοδότηση από τα περιθώρια της γραμμής 4 του τη συμφωνία Πλαισίου ή από άλλες δυνατότητες από το Δημοσιονομικό Πλαίσιο Εξωτερικών Δράσεων όπως τα ευέλικτα μέσα. Ευχαριστώ πολύ. Bene. Mm, l'onorevole Galler è stato Ο κύριος Γκάλερ ήταν εισηγητής στην προηγούμενη θητεία σχετικά με το μέσο συνεργασίας και ανάπτυξης. Δικαιούται λοιπόν να λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από χτες το σχέδιο έκθεσης πλέον ε, διατίθεται και το εξετάζω λοιπόν. Από χτες δεν μπορώ να τοποθετηθώ οριστικά αλλά θεωρώ ότι η συνεργασία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Εσωτερικών Υποθέσεων και της δική μας Επιτροπής, παρά το γεγονός ότι είμαστε συνδεδεμένες, ε, θα μπορούσε να είναι καλύτερη και νομίζω ότι αυτό θα διευκολύνει και το έργο της εισηγήτριας. Σκοπός της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως είπε, είναι να γευρεωθεί ένα χάσμα σε ένα τέτοιο μέσο εξωτερική πολιτικής. Επειδή είναι πολύ περιορισμένη ο συντονισμός ε, του μέσου ανάπτυξης και έτσι δεν διευκολύνονται τα μέτρα τα οποία προβλέπονται μετά την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας και μετά την εμφάνιση του προβλήματος της νομικής βάσης, φαίνεται ότι επικρατεί μια νέα συνένεση προς την κατεύθυνση αυτή και ευχαριστώ την εισηγήτρια για την υποστήριξη του συμβιβασμού σε ό,τι αφορά τη νομική βάση, βάση τη, λόγω της μεγάλης γεωγραφικής έκτασης που καλύπτεται και των χρηματοδοτικών μέσων, μέσων αναφέρθηκε αυτό άλλο, άλλωστε, προβλέπεται επέκταση των μέσων και αναφέρεται επέκταση κατά 176 εκατομμύρια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να συμπεριληφθεί και να χρηματοδοτηθεί εν μέρη το ε, ποσό αυτό από τον DCI. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ περιορισμένο το ποσοστό αυτό και ότι θα πρέπει τα μέσα να ανταποκρίνονται και στις εργασίες, στα καθήκοντά μας για την επιτροπολογία τώρα. Η Επιτροπή μας τους κοιόδες και τους ε, βασικούς εισηγητές στους έδωσε το Δεκέμβριο την εντολή να ξεκινήσουν διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξασφαλίσουμε την μεγαλύτερη δυνατή επιρροή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της Επιτροπολογίας. Θα ήθελα να ζητήσω σήμερα ξανά τα άτομα αυτά να συμμετάσχουν πραγματικά στις εργασίες, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι ουσιαστική η συμμετοχή τους. Επίσης μου έκανε εντύπωση μία λεπτομέρεια στο κείμενο. Το μέσο γεωγραφικά θα εφαρμοστεί και στη Μέση Ανατολή και υπάρχουν πολλές ε, περιοχές οι οποίες αναφέρονται και με συνδημογραφίες. Και βρήκαμε μια συνδημογραφία η οποία αναφέρεται αμάς. Σε κάποιες γλώσσες, όπως ξέρετε, το χα της χαμάς δεν προφέρεται. Άρα το αμάς και χαμάς θα ακούγεται το ίδιο, ταυτόσιμο. Ίσως λοιπόν θα μπορούσαμε κάπως να αλλάξουμε τη σειρά των αρχικών για να μην αναφέρεται ως μέσο συνεργασίας το άμα στη Μέση Ανατολή. Να το πούμε σάμα, να το πούμε κάπως αλλιώς τέλος πάντων, όχι αμάς. Ενδιαφέρουσα αυτή η παρατήρηση ε, σας ε, για το ακρονίμιο. Ο κύριος Αλαφράγκα. Ευχαριστώ. Πέραν της ε, πολεμικής που μπορεί να προκαλέσει η χρήση κάποιων ακρονιμίων, ε, θα θέλω να πω ότι μόλις λάβαμε το έγγραφο, εγώ εντάχει το διέτρεξα, ε, και το κείμενο δεν είναι πλήρες διότι δεν περιέχει τα παραρτήματα και ειδικά το παράρτημα 2 που είναι το ουσιοδέστερο που αναφέρεται ο κατάλογος των χωρών στις οποίες κατανέμονται τα κονδύλια. Λοιπόν, ε, ένα από τα βασικά ζητήματα που έχει το θέμα αυτό είναι η νομική βάση και η συγκήτρια προσπάθησε να εμπλέξει, να μίξει το κοινοβούλιο σε αυτή τη διαδικασία. Με το κοινοβούλιο πρέπει να επιμείνει σχετικά με τη συγκεκριμένη εφαρμογή τη νομική βάση, όπω προτείνει η συγκήτρια μετά από τη θέση ισχύ τη συνθήκη τη Αβώνα τώρα. άλλο ζήτημα κατά πόσον η αύξηση των πόρων επαρκεί ε, σε σχέση με την αύξηση των χωρών που θα απολάβουν ε, αυτά τα ωφέλη από την πρωτοβουλία θα πρέπει να το επανεξετάσουμε όπως επίσης και την κατανομή που προτείνει η Κομισιόν. Να ζητήσω από την εισηγήτρια ποια είναι η ε, άποψή της σχετικά με την πρικοδότηση που προτείνει η Κομισιόν, αν είναι ικανοποιητική, αν επαρκεί απέναντι στις υποχρεώσεις που ανταλαμβάνουμε μέσω του κανονισμού. Ε, κάτι ακόμα πρόεδρο, δεν ξέρω ποια θα είναι η τελική διαδικασία, αλλά τώρα που η Επιτροπή μας θα έχει αυτή τη γνωμοδότηση, εμείς θα ενεργήσουμε βάσει τον ε, άρθρο 50 σε ό,τι αφορά την ε, συνεργασία με άλλη επιτροπή, αλλά νομίζω ότι εμείς μπορούμε να βάσει τον αρμοδιοτήρο μας να δραματίσουμε έναν ρόλο πολύ πιο ενεργό και να παίξουμε ένα ρόλο που θα μας βοηθήσει μαζί με τις άλλες επιτροπές να προαγάγουμε ιδιαίτερα αυτό το μέσο. Ε, να σας απαντήσω κύριε Σαλαφράνκα. Σκεφτήκαμε από εκείνο με την νομική υπηρεσία να εφαρμόσουμε το άρθρο 50 όπως είπατε και εσείς σε αυτή την περίπτωση. Ισχύουν λοιπόν τα γενικά κριτήρια ως εκ τούτου εμείς είμαστε καταρχάς ε, αρμόδιοι και υπεύθυνοι αλλά σε συνεργασία με άλλες επιτροπές. Το λόγο έχει ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρία Μίλλερ. Ε, thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως και κάποια άλλα κάποιοι βουλευτέ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε το κείμενο αυτό χθε μόλι. Την εξετάσαμε λοιπόν με προσοχή, αλλά δεν μπορούμε ακόμα να τοποθετηθούμε οριστικά σήμερα. Δύο γενικέ παρατηρήσει θα ήθελα να κάνω όμω. Καταρχά για το χρονοδιάγραμμα και κατά δεύτερον για το θέμα τη επιτροπολογία, το οποίο το έθιξε και η Επιτροπή σα. Γενικά, όπως είπε ο κύριος Γκάλερ, σκοπός της πρότασής μας ήταν να πληρώσουμε χάσμα που υπήρχε στην νομοθεσία. Και τι εννοούμε, ότι υπήρχαν κάποια προγράμματα τα οποία όλα θέλουμε να χρηματοδοτούνται στις χώρες εταίρους, αλλά δεν μπορούμε να τα χρηματοδοτήσουμε μέσω του μέσου ανάπτυξης και συνεργασίας. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν έναν τρόπο να ε, γεμίσουμε κάπως να, αυτό το κενό που υπήρχε. Διατίθενται λοιπόν τα κονδύλια αυτά στο προπολογισμό αυτό και θα πρέπει να προσαρμοστεί η πρόταση αυτή το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να χορηγηθούν τα κονδύλια αυτά από τον τρέχοντα προϋπολογισμό. Ανησυχούμε κάπως σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζουμε να βοηθήσουμε και να επιταχυνθούν οι εργασίες στην Επιτροπή ΑΦΕΤ. Θα θέλαμε να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο την κυρία Λόχ Μπίλτερ και τους υπόλοιπους βουλευτές για να καταλήξει σε μια οριστική θέση το θέμα αυτό και θα πρέπει να δούμε αν τα καταφέρουμε να συμφωνήσουμε. Για το θέμα της επιτροπολογίας, ε, Πρόεδρε, έχουμε δηλώσει και στο παρελθόν ποια είναι η άποψή μας ενώπιον της Επιτροπής σας. Το Συμβούλιο θα κοινοποιήσει τη θέση του στις τριμερείς συνομιλίες οι οποίες διοργανώνονται στην παρούσα φάση. Άρα θεωρώ ότι θα υπάρξει σχετικό τριμερής διάλογος μεταξύ των τριών ε, οργάνων και προφανώς τίθεται θέμα διαφορών ως προς την νομική ερμηνεία για τη νέα συνθήκη, αλλά να επαναλάβω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να βρεθεί λύση για το θέμα αυτό και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια εκ μέρους μας για να βρεθεί όντω μία λύση, να διευκολυνθεί μία συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Θα αντιδραματίσουμε ενεργό ρόλο λοιπόν στις τριμερείς αυτούς διαλόγους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Και τώρα μπορούμε να κλείσουμε νομίζω τη συζήτηση. 10 Φεβρουαρίου του 2010 στις 6 έχουμε την προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών και τελική εξέταση με ψηφοφορία στην Επιτροπή μας στις 17 Μαρτίου. Θα διακόψουμε για πολύ λίγο, γιατί είμαστε μπροστά, σχέση με το πρόγραμμα κατά 6 λεπτά. Α, η κυρία Λόκμπίλερ. Ναι, θα σας ε, ακούσουμε αξιοποιώντας αυτά τα 6 λεπτά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ίσως να μην χρειαστούν και τα 6 λεπτά. Στο συγγνώμη ε, που είχαμε τόσο μικρό χρονικό περιθώριο. Είπε και ο κύριος Αλαφράνκα ότι λείπει το παράρτημα και εγώ είμαι διατεθειμένη βεβαίως πάντοτε να ακούω τις παρατηρήσεις και υποδείξεις για τα διάφορα θέματα και να τη μαζί σας. Ρωτάει ο κύριος Σαλαφράνκα πώς ε, βλέπω εγώ αυτή την κατανομή των κονδυλίων. Κοιτάξτε, καταρχάς έχουμε να κάνουμε ένα πρώτο βήμα. Η Επιτροπή μέχρι στιγμή έχει χειριστεί την υπόθεση κατά 50-50%. Εμεί θα προτείναμε να μετατοπιστεί το βάρο και να πάμε στα 2 τρίτα, 1 τρίτο, αλλά βεβαίω να ακούσουμε τι έχει συγκεκριμένα να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναλόγω να κάνουμε τι διευκρινήσει. Για τον κύριο Κάλλερ, η ε, συμμετοχή στο δρυμερή διάλογο που ξεκινάει το Φεβρουάριο βεβαίως και θα συμπεριλάβει και εμάς, θα είμαι και εγώ παρούσα, θα ήθελα να συμπληρώσω επιπλέον ότι το μέσον αυτό δεν περιλαμβάνει τη Μέση Ανατολή. Αν έχετε όμως, ε, και ως εκ τούτου θα πρέπει να υπάρχει πρόβλημα προς το ακρονίμιό του, αν όμως έχετε κάποια διαφορετική ιδέα, πολύ ευχαρίστως να την ακούσουμε. Ε, επίσης θέλω να πω ότι το χρονοδιάγραμμα ξέρω ότι είναι ε, στενό, πιεστικό, αλλά ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να το τηρήσουμε και θα ήταν καλό να ακούσουμε, ε, να έχουμε την ευκαιρία να ψηφίσουμε μέσα στην Επιτροπή μας στις 23 ακόμη Φεβρουαρίου για να προλάβουμε άλλες προθεσμίες. Ευχαριστώ. Πολύ καλή η πρότασή σας και εύχομαι να μπορέσει να υλοποιηθεί η σκέψη σας. Λοιπόν, ένα διαλυματάκι πεντάλεπτο για να ξεκινήσουμε μετά σε 11 και ακριβώς. Αν φτάσει ο κύριος Τόμας Ντούπλα, για να περάσουμε στο επόμενο σημείο και τελευταίο για σήμερα το πρωί.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 Bene, cari colleghi, possiamo iniziare l'ultimo punto all'ordine del giorno. ανταλλαγή απόψε με την Επιτροπή. Το προσωπείται από τον διευθυντή που είναι υπεύθυνο για τη συνεργασία με τις μεσογειακές χώρες, ο κύριος Δεμοράλ για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των μεσογειακών χωρών για την περίοδο 2011-2013. Όπως ξέρετε σήμερα η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει δύο συζητήσεις για την στρατηγική γειτονία, καταρχάς ό,τι αφορά τις μεσογειακές χώρες. Αυτή η συζήτηση θα ξεκινήσει τώρα. Και η άλλη συζήτηση για την ανατολική εταιρική σχέση. Θα ξεκινήσει σήμερα το απόγευμα. Σημαντικό νομίζω είναι να κάνουμε κάποια εισαγωγικά σχόλια. Σήμερα το θέμα δεν είναι να συζητήσουμε απλά πολιτικές προτεραιότητες. Η πολιτική γειτονία, από ό,τι ξέρετε, βασίζεται σε ένα πρόγραμμα χρηματοοικονομικής ενίσχυσης και το εργαλείο του σχετικό, αλλά και οι διαδικασίες εφαρμογής συνοδεύονται από διαβουλεύσεις και από στενό διάλογο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των χωρών που α, χρησιμοποιούν την βοήθεια αυτή. Από το 2007, όταν το εργαλείο κατέστη πλήρως λειτουργικό, η Επιτροπή μας ζητούσε διαρκώς το δικαίωμα παρακολούθησης και καθοδήγησης του τρόπου κατά τον οποίο ταπανώνται τα κοινωτικά κονδύλια προς τις χώρες αυτές. Πρόκειται για ένα ρόλο που αρμόζει σε μια κοινοβουλευτική συνέλευση, αρμόζει σε εμάς. Για να εξηγήσουμε τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες θα καθοδηγήσουν την ε, κοινοτική ενίσχυση τα επόμενα χρόνια και για να λεφθεί υπόψη και η δική μας θέση. Έχουμε εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μαζί μας εδώ σήμερα. Λάβατε επίσης αναλύσεις, επισκοπήσεις, συνοπτικά στοιχεία τα οποία έχουν καταρτήσει εμπειρογνώμονες, τα οποία θα σας βοηθήσουν κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Σας τα διαβίβασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να δώσω λοιπόν το λόγο τώρα στον κύριο Τόμας Ντούπλερ Μοράλ για την εισαγωγή του. Και μετά οι συνάδελφοι θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις, να κάνουν σχόλια για να αρχίσει ο διάλογος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το λόγο λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Όπως ευχαριστώ και τη γραμματεία που διοργάνωσε τόσο γρήγορα τη συνάντηση αυτή για την ε, ταχεία ανάλυση των στρατηγικών εγγράφων και των ενδεικτικών προγραμμάτων αναχώρα. Και χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ για την ανταλλαγή αυτή απόψεων σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αναθεώρησης για την ε, στρατηγική αυτή και όπως είπατε ε, θα χαρώ να είναι ανοιχτός ο διάλογος και στενός με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν χρειάζεται να σας αναφέρω γιατί η Μεσογειακή περιοχή είναι σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που συνεπάγεται η περιοχή αυτή για εμάς, αλλά και σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες καταπολέμησης και σταθεροποίησης της ευρύτερη περιοχή. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχει η περιοχή. Δεν έχουμε δικαίωμα να είμαστε απόντες. Θα πρέπει με την πολιτική μας να προωθήσουμε τις ευρωπαϊκές αρχές και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία παραμένει το γενικό πλαίσιο πολιτικής σε ό,τι αφορά την περιφερειακή συνεργασία. Ξέρετε ότι η Αλγερία, η Συρία και η Λιβύη είναι χώρες που δεν έχουν ακόμα ενσωματωθεί πλήρως και έχουμε ξεκινήσει ε, στην Αίγυπτο και σε άλλες χώρες επιτυχεί προγράμματα και έχουμε διάφορους εταίρους που ε, συμμετέχουν ενεργά στην πολιτική αυτή. Όπως ξέρετε, η πολιτική κατάσταση στην περιοχή, στις περισσότερες από τις χώρες αυτές, είναι σταθερή. Φυσικά υπήρχαν σημαντικές εξαιρέσεις, όπως για παράδειγμα ότι ακολούθησε την σύγκρουση τη Γάζα ή την πολιτική δήλωση το Λίβανον. Έγιναν εκλογές σε πολλές χώρες, αλλά οι οποίες δεν επέφεραν αλλαγή των κυβερνητικών σχημάτων. Και ενώ συνεχίζεται η διαδικασία, δεν μπορούμε να πούμε ότι συνεχίζεται και ο εκδημοκρατισμός σε ό,τι αφορά θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατικής διακυβέρνησης. Είναι περιορισμένη η πρόοδος. Ωστόσο, συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας στην περιοχή αυτή και ο διάλογος έχει εντατικοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, αποστείλουμε ε, παρατηρητικές εκλογές για τις εκλογές, ε, ε, αποστολές για την εκλογές στο Λίβανο και επίσης στην Αίγυπτο, την Ιορδανία, το Μαρόκο, την Ισία και στην Αλγερία συμφωνήθηκε πρόσφατα να οικοδομηθούν δομές τέτοιου διαλόγου. Οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις έχουν λάβει μια όθηση και χάρη στην υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η την Ισία και ο Λίβανος έχουν λάβει ενίσχυση για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η Αίγυπτος ε, έχει αναλάβει προγράμματα για θέματα απελευθέρωσης της αγοράς και οικονομικής συνεργασίας. Νομίζουμε ότι ο διάλογος και η συνεργασία με όλες αυτές τις περιοχές καθώς και η υποστήριξη από τα μέσα συγκεκριμένων μέσων αποφέρει καρπούς ε, στις μεσογειακές χώρες. Για παράδειγμα, το Μαρόκο και η Αίγυπτος αποτελούν τις πρώτες χώρες ε, απορρόφησης των κινητικών προγραμμάτων στο Μαρόκο ε, υπάρχουν 45 προγράμματα και η Αίγυπτος αποφαλείται από 30 και πλέον τέτοια προγράμματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ο βασικός επενδυτής και εταίρος των χωρών αυτών για χώρες όπως ο Λίβανος και η Ιορδανία και είναι διψήφια τα ποσοστά πλέον από το 2008 και εξής. Επίσης, έχουμε αυξήσει τις εμπορικές ροές. Το 2008 αυξήθηκαν ε, οι εμπορικές σχέσεις με το Λίβανο και σε ό,τι αφορά τομείς όπως η γεωργία και οι δημόσιες υπηρεσίες έχουμε ξεκινήσει ε, πολλές διαπραγματεύσεις σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση του εμπορίου θα αποτελέσει ένα κλειδί για την οικονομική εξυγχρονισμό των εταίρων μας, δίνοντας ευκαιρίες και στην ύπεθρο. Αυτό θα περιορίσει την πίεση και την αστεφιλία και τις κινήσεις της μεταυστατικής προς την Ένωση. Η προσέγγιση τους γενικά είναι πιο συντηρητική σε ό,τι αφορά τα εμπορικά, τα σύγχρονα εμπορικά σχήματα, ωστόσο ε, τους έχει χτυπήσει η κρίση η οικονομική της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τις μείωση των επενδύσεων και του τουρισμού. Πολλές χώρες ζήτησαν ενίσχυση της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί θεωρούν να αποτελεί αυτό ένα κλειδί για τον οικονομικό τους εξυγχρονισμό. Η συμφωνία για προηγμένο καθεστώς στο Μαρόκο που συνήφθη το 2008 προλύανε το έδαφος για τις καλύτερες διμερείς σχέσεις μέσω της ε, ιδιαίτερης συμμετοχής των θεσμών αφότρων των χωρών και εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι δημιουργήθηκε μια κοινή κοινοβουλευτική επιτροπή που εγκρίθηκε πρόσφατα από το Μαρόκο αλλά και με την ΕΟΚΕ και με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η συνεργασία μας με την Ορδανία και την Αίγυπτο ενισχύθηκε και έτσι και οι δύο χώρες πλέον θέλουν να αναβαθμίσουν τις σχέσεις τους με την Ένωση. Και το ίδιο ισχύει και για την Τινησία. Οι διαπραγματεύσεις για την σχέσεις, ε, σχέσεις με τη Σύρια επανακινήθηκαν από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να ολοκληρώσει τη συμφωνία αυτή. Τώρα η Συρία θέλει να εκτιμήσει θέλει περισσότερο χρόνο για να εκτιμήσει τον οικονομικό αντίκτυπο στις χώρες και ενδεχομένως να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς σχέσεις. Σε ό,τι αφορά τη Λιβύη, τον Νοέμβριο του 2008 ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις οι οποίες και βρίσκονται σε συνέχιση με την Αλγερία. Συμφωνήσαμε επί ενός οδικού χάρτη, ο οποίος θα δώσει νέα όθηση στις σχέσεις μας και την επόμενη εβδομάδα θα παρευρεθώ και εγώ στην Αλγερία για να δώσω ακριβώς περαιτέρω όθηση στις διαπραγματεύσεις στο μέσο αυτό. Η ανάπτυξη της πολυμερούς πτυχής ε, της μεσογειακής ε, περιοχής ενισχύθηκε το 2008 που όπως ξέρετε σκοπό η σύνοδος αυτή είχε να αναβαθμίσει το πολυμερές επίπεδο. Δημιουργώντας και μια σχεδιακή γραμματεία και γραφεία ενημέρωσης στις χώρες αυτές για να βλέπουν οι πολίτες ποιος είναι ο συγκεκριμένος αντίκτυπος. Από την συνάντηση στη Μασαλία πέρσι έγιναν κάποιες πρόοδοι σε ό,τι αφορά την ίδρυση του σχετικού γραφείου στην Βαρκελόνη. Και θα πρέπει φυσικά να δούμε ποια είναι τα προγράμματα προτεραιότητας. Όπως ξέρετε, οι εξελίξεις και η πρόοδος ε, παρακολύεται από τις ε, συγκρούσεις στην Μεσανατολή ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα, τις συγκρούσεις στη Γάζα το 2008. Είναι πολύ υψηλό το επίπεδο της φιλοδοξίας των εταίρων μας, αλλά γενικά επικυρώνεται η στρατηγική μέθοδος την οποία επιλέξαμε πριν από, κάποιες, από κάποια χρόνια και προφανώς ε, έχει προσαρμοστεί το πεδίο των προτεραιοτήτων μας ε, τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει να προχωρήσουμε τις προσπάθειες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη Λιβύη και τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Για τη Λιβύη, οι συζητήσεις και διαβουλεύσεις ε, μας έδωσαν ένα πολιετές πρόγραμμα. Δυστυχώς για την Παλαιστινιακή Αρχή δεν μπορεί να γίνει πολιετές προγραμματισμός σε αυτή τη φάση λόγω της κατάστασης. πρέπει να έχουμε μια συνεκτική προσέγγιση για όλα τα προβλήματα στην Μεσόγειο και θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τις νέες εξελίξεις στην περιοχή προκειμένου στους στόχους του 2011 και 2013 να εντοπίσουμε νέες προτεραιότητες και θα έχουμε και πιο πολλά κονδύλια. Το 2010 ε, ο προπολογισμό ήταν 850 εκατομμύρια για κάθε χώρα. Το 2012 θα είναι ένα δις το ποσό αυτό. Και ιδιαίτερα μέσω του ε, μέσω ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Όλα αυτά θα αποστέλουν ένα μήνυμα προς τις χώρες αυτές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διατίθεται να τις βοηθήσει και να τις ε, ενισχύσει. Θεωρούμε ότι υπάρχει σωστή ισορροπία σε ό,τι αφορά την εκχώρηση πόρων. Η πιο υψηλή εκχώρηση είναι προς το Μαρόκο. Δεύτερη είναι η Αίγυπτος και αυτό αντικατοπτρίζει την στρατηγική της συμφωνία. Η Ορδανία λαμβάνει υψηλά κονδύλια κατά κεφαλή και είναι ανάλογη και η δέσμευσή της για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την ε, γειτονία. Αναφερθήκατε στις διαβουλεύσεις που έγιναν. Όντως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μια συμμετοχική μέθοδο προσέγγισης και διοργάνωσε μια ευρεία διαβούλευση όπου συμμετείχαν και οι τοπικοί αλλά και οι διεθνείς εμπλεκόμενοι φορείς. Αυτό επιτρέπει και στην κοινωνία των πολιτών να σχολιάσει την προσέγγιση που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπου ήταν δυνατόν αυτόν, ε, γεωγραφικά, ε, τοπικές μάλλον υπηρεσίες, διοργάνωσαν μία τοπική ε, συνάντηση με τα εμπλεκόμενα μέρη αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν τοπικές εκπροσωπήσεις μέσω της ε, Επιτροπής των Βρυξελών. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα για τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αναθεώρησης. Στο Λίβανο προτείναμε να αναπτυχθούν ε, διάφορες πολιτικές ό,τι αφορά την, ε, το περιβάλλον. Στην Ιορδανία θέλουμε να καταπολεμήσουμε την αλλαγή του κλίματος, βελτιώνοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα και επίσης υποστηρίζουμε τη μεταρρύθμιση της, ε, των δημόσιων υπηρεσιών στην Αίγυπτο. Θα υποστηρίξουμε μακροπρόθεσμες ε, προοπτικές ανάπτυξης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αλλαγή του κλίματος, για την ενίσχυση ε, της ενεργειακής αποδοτικότητας. Στο Ισραήλ θα βοηθήσουμε το σχέδιο, την εφαρμογή του σχεδίου δράσης σε ό,τι αφορά τη ε, συνεργασία μεταξύ των θεσμών στον Μαρόκο, αποφασίσαμε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση των διαθεσμικών ε, ικανοτήτων και του συντονισμού με τα ευρωπαϊκά πρότυπα στην Αλγερία και στην Τινησία. Θα εστιαστούμε βασικά σε οικονομικό εξυγχρονισμό, αλλά θα εστιαστούμε στο κλίμα και στο περιβάλλον αλλά και σε θέματα ανάπτυξης υπέτρου και της γεωργίας για να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να κινητοποιηθεί η μικροπιστωτική βοήθεια προς τις χώρες αυτές. Αυτό ευτυχώς δεν χρειάζεται επί του παρόντος για τις χώρες αυτές. Προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τα επενδυτικά μέτρα τα οποία θα ενισχύσουν την ανάπτυξη και έχουν αυξηθεί σημαντικά οι εκχωρήσεις για την περίοδο 2011-2013. Επίσης ε, αυξήθηκαν οι δανεισμοί της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και μπορεί να αυξηθούν και περαιτέρω. Τέλος, σε ό,τι αφορά την περιφερειακή συνεργασία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε για την περίοδο 2009-2010 επιπλέον 70 εκατομμύρια τα οποία θα καταπολεμήσουν την ρήπανση στη Μεσόγειο, θέματα εκπαίδευσης και έρευνας. Ε, συγγνώμη, αλλά με ενημέρωσαν οι διερμηνείς ότι διαβάζεται με ιδιαίτερα υψηλή ταχύτητα. Ε, Παρακαλώ, ο καιρός θα ήταν ε, χαμηλός σε ταχύτητα. Ευχαριστώ. Δεν ήθελα να σας απασχολήσω για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά καταλαβαίνω τι λέτε. Αυτό που έλεγα είναι ότι για την περιφερειακή συνεργασία, πέρα από τα 70 επιπλέον εκατομμύρια που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2009 να χορηγήσει, προφανώς θα υπάρξει μέσω προγραμματισμού για την περιοχή αυτή, το οποίο θα επανεξεταστεί χρόνο. Ελπίζω να κατάφερα να σας παρουσιάσω ποια ήταν η εξέλιξη των σχέσεών μας με τους ε, εταίρους μας της μεσογειακών χωρών. Ίσως να μίλησα πάρα πολύ γρήγορα, αλλά αναφέρθηκα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και στο πώς προγραμματίζουμε να τις βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και όπως είπα στην αρχή θα χαρώ να γίνει διάλογος για όλα αυτά τα θέματα. Eh, eh, Και τώρα θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Η κυρία Φλότρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση στη Μεσόγειο εντάσσεται σε ένα πλαίσιο το οποίο προέκυψε από τη δικασία τη Λισαβόνα και νομίζω ότι η δυσκολία που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι να συνοδεύσουμε την λόγω διαδικασία η οποία παρατηρούμε ότι υλοποιείται σε ενισχυμένο στάδιο, δηλαδή για ένα πολιτικό διάλογο, οικονομική ενίσχυση κλπ. να τον υλοποιήσουμε αναφορικά με τα κριτήρια της Κοπενχάγης για θέματα διεύνησης. Δηλαδή έχουμε ανάγκη από ένα είδος ε, κριτηρίων τα οποία θα εφαρμόζονται, θα είναι γνωστά στα κράτη με τα οποία συζητάμε και τα οποία χρηματοδοτούν μια σειρά προγραμμάτων και αυτοί θα είναι οι στόχοι που θα μας καθοδηγούν παντού και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Νομίζω ότι αναφέρεται ρητά, αν δεν κάνω λάθος, σε αρκετά έγγραφα αξιολόγησης που μας υποβάλλατε ότι η οικονομική, η δημοσιονομική και εμπορική πτυχή δεν μπορεί να προχωρήσει Παραδείγματο χάρη, αν η ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη δεν προχωράει παράλληλα, η καταπολέμηση τη διαφθορά δεν βρίσκεται στον πυρήνα του προγραμμάτων. Φυσικά χρειάζεται ευελιξία. Κάθε χώρα δεν έχει η μία κατάσταση σε μια χώρα δεν είναι ίδια με αυτή που επικρατεί σε μια άλλη, δεν υπάρχουν τα ίδια μέσα και λοιπά. Υπάρχει, δεν υπάρχει διαβούληση, αλλά θα πρέπει στην Μεσόγειο να έχουμε σαφή κριτήρια και δεν θεωρώ ότι μπορούμε για οποιαδήποτε από αυτές τις χώρες να παραβλέψουμε την χρηστή διακυβέρνηση, την καταπολέμηση δικαιοσύνη, την ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα που θα πρέπει να παραμείνουν στον πυρήνα της όλης υπόθεσης. Γνωρίζουμε εξάλλου ότι όλα τα θεώσεις αυτές τις χώρες ε, προσπαθούμε να τις κινητοποιήσουμε για να καταπολεμήσουν την παράνομη μετανάστευση, να τους ζητήσουμε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Θεωρώ λοιπόν πως χρειάζεται να αποδώσουμε ιδιαίτερη προσοχή πάνω στο θέμα. Καμία από τις χώρες δεν έχει ένα αποτελεσματικό δικαίωμα ασύλου που θα προστατεύει όλες τις χώρες αυτές. Ε, το θέμα της ε, εξόδου από την χώρα, ο καθένας έχει το δικαίωμα, αλλά αυτό δεν συμβαίνει στις περιπτώσεις αυτές. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα ήθελα να ε, βρίσκονται συστηματικά στις ε, σχέσεις μας και στις εκθέσεις με τις χώρες αυτές και δεν βλέπω να συμβαίνει. Τώρα, το παράδειγμα της Τινησίας, διότι το συζητήσαμε την περασμένη εβδομάδα και ολοκληρώνω εδώ, το ζητήσαμε στο Λομέλια λοιπόν, διότι κάνετε μια ανάλυση που εντάξει δεν είναι κακή. Λέτε πως εάν οι βάσει για μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη είναι, στηρίζονται στην, στο Σύνταγμα, αλλά τόσο το Ανώτατο Δικαστήριο όσο και η εισαγγελία ελέγχονται από την εκτελεστική εξουσία. Όταν διαβάζει λοιπόν κανείς αυτή την ανάλυση που βρίσκονται στο επίκεντρο του σχεδίου ε, συνεργασίας με την Τινησία και λέμε ότι αυτό είναι το ενδεικτικό πρόγραμμα για τις χρονιές, θα πρέπει να στηριχθούμε σε ένα στόχο που θα αφορά στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στην Τινησία. Διαβάστε λοιπόν αυτό το ενδεικτικό πρόγραμμα της Τινησίας και θα δείτε ότι δεν υπάρχει ούτε μια κουβέντα πάνω σε αυτό. Ακόμα και τα κριτήρια αξιολόγηση της δικαιοσύνης δεν αναφέρονται στο δικαστικό σύστημα της Τινησίας που βρίσκεται ουσιαστικά στα χέρια του Προέδρου και του κόμματος ε, που κυβερνά. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν ποια μπορεί να είναι τα μέσα και πρέπει να είναι τα μέσα μιας ε, δικαιοσύνη ε, που αναφέρονται σε ένα ενεργητικό πρόγραμμα, ακόμα και αν η ανεξαρτησία της δεν είναι καν στόχος αυτής της προσπάθειας. Υπάρχουν λοιπόν <clears throat> διάφορες ασυνέπειες, αλλά όπως σας είπα και πριν, αυτό συμβαίνει σε κάθε χώρα. Φυσικά αυτές οι συνέπειες είναι διαφορετικές από χώρα σε χώρα. Και θα μου πείτε ότι δεν θέλουν καν να το ακούσουν και αν τους μιλήσουμε για ανεξαρτή δικαιοσύνη θα μας πούνε γεια σας. Το προχωρημένο ε, καθεστώς σημαίνει ενισχυμένη συνεργασία, δηλαδή συμφωνία σε θεμελιώδεις αρχές που αφορούν στις σχέσεις μας με τις μεσογειακές χώρες. Αυτό δεν συμβαίνει με την περίπτωση της Τινησίας, αλλά έχω και άλλα παραδείγματα, δεν θέλω να μακρηγορήσω. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα, ελπίζω ότι οι συνάδελφοι θα τα θίξουν, όπως π.χ. το Ισραήλ και άλλα που δεν μας ικανοποιούν διόλου σε ό,τι αφορά τους στόχους μας όπως έτυχαν διαπραγμάτευσης. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω κάποιες ερωτήσεις προς την Επιτροπή σχετικές με τη Συρία. Γνωρίζετε ότι η υπογραφή της ε, συνθήκης ε, συνεργασίας με την Συρία, μεταξύ Συρίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σε εκκρεμότητα, και όμως αποτελεί μια προϋπόθεση έτσι ώστε να ε, εξασφαλιστεί ένα σαφές πλαίσιο για αυτή την πολιτική γειτονίας. Και γι' αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στις προτεραιότητες του Εθνικού Προγράμματος 2011-2013, οι οποίες δεν είναι σαφείς. Όλα αυτά θα έπρεπε να είναι λεπτομερέστερα. Και στο πλαίσιο αυτό ζητώ από την Επιτροπή να μας πει τι στρατηγική σκοπεύει να ακολουθήσει έναντι της Συρίας. Έχει κάποιο άλλο ε, σχέδιο υπόψη κάποια εναλλακτική σε περίπτωση που δεν ε, υπογράψει συμφωνία ε, συνεργασία στη Συρία. Επίση, σε σχέση με τα όσα είπε η κυρία Φλότρο για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνη το δικαστικό σύστημα κτλ. Το ενδεικτικό πρόγραμμα της Συρίας δεν είναι βιώσιμο με αυτές τις συνθήκες και θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες από την Επιτροπή. Επίσης, προς την ενίσχυση του ρόλου της Κοινωνία των πολιτών που έχει εγγραφεί μέσα στο αντικείμενο του νέου προγράμματος ως στόχος εξέλιξης ε, ανάπτυξης της Συρίας. Ρωτώ λοιπόν, θα μπορούσαν ζητήματα ανθρωπινών δικαιωμάτων να ενσωματωθούν στα προγράμματα τα σχετικά με την κοινωνία των πολιτών, τουλάχιστον ω προ τα κοινωνικο-οικονομικά δικαιώματα. Ευχαριστώ. Μάιερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα την επιχειρηματολογία της κυρία Φλόιου. Είναι γεγονός ότι η πολιτική γειτονία ε, που υποστήριζε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η πολιτική ε, επηρέαζε τις, ε, μάλλον συνδυάζει τις εξελίξεις στις ε, γειτονικέ χώρες με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ε, ελευθερία. Το άρθρο 2 λοιπόν αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρηθούν αυτοί οι κανόνες. Νομίζω ότι αυτό το ζήτημα τώρα πια δεν λαμβάνεται και τόσο πολύ υπόψη τουλάχιστον στην Μεσογείο. Μεσογείου. Υπάρχουν δύο χώρες που είναι υποδειγματικές ε, σε ό,τι αφορά την ε, <clears throat> απάρνηση εφαρμογής αυτού του άρθρου 2, το Μαρόκο και το Ισραήλ. Το Μαρόκο το Μάρτιο και μάλλον ε, το Μαρόκο έχει αποκτήσει το καθεστώς της πλέον ευνούμενης χώρας συνεχίζει να κατέχει την περιοχή της Δυτικής Ζαχάρας, να καταπιέζει τους πολίτες ε, της Δυτικής Ζαχάρας ε, συστηματικά και παραμελεί και παραβιάζει συνεχώ και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Σε μια, υπάρχει και μια αποστολή της Μινούρσου των Ηνωμένων και τελευταία στον Μαρόκο και στα κατεχόμενα εδάφη υπάρχει καταπίεση των πολιτών. Παράδειγμα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, είναι το, ίδιο μια χώρα όπως το Μαρόκο ή το Ισραήλ να παραβιάζουν, μιλάμε το, για το Ισραήλ στην περίπτωση της ε, Γάζας, ε, παραβιάζοντας ε, το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις, για μας δηλαδή είναι το ίδιο. Είτε μια χώρα ε, πληρεί τις προϋποθέσεις είτε όχι, εάν σέβεται τα δικαιώματα είτε όχι. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποκατασταθεί και αυτό το μέσο γειτονίας να μπορεί να εφαρμοστεί μόνο στις περιπτώσεις που δεν γίνονται τέτοιε ε, παραβιάσεις υπάρχει μια κόκκινη γραμμή. Για αυτή την μάλιστα την ανέφερε και το Ισραήλ, δηλαδή για την ε, σύσταση δύο κρατών, ε, ανεξαρτήτων κλπ. Υπήρχαν λοιπόν κάποιες συμφωνίες και τελικά δεν έγινε τίποτα και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως απάντηση τι έγινε. Σφυρίζει αδιάφορα. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν ότι δεν υπάρχει μια ε, σωστή εφαρμογή αυτού του μέσου γειτονία. Δεν μπορεί λοιπόν να διαφορεί ε, σε συμπεριφορές όπως αυτές του Ισραήλ και του Μαρόκου. Το Συμβούλιο της Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών έχει προτείνει την διαδικασία από απεικιοποίησης που εκρεμεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση που ήταν χώρες απειγιοκρατικές θα έπρεπε τουλάχιστον να έχουν την ελάχιστη εδώ και μπροστά σε τρίτε διαδικασίες από να απαιτήσουν από το Μαρόκο να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο από Και η Κομισιόν όταν μιλάει και θίγει το ζήτημα των ε, χρηματοδότησης και βοήθειας προς το Μαρόκο, αναφέρει ότι ε, παρήχε βοήθεια σε προγράμματα που υποστηρίζουν τη διαχωρισμό των ε, αρμοδιοτήτων, των εξουσιών, αλλά αναφέρεται ότι αυτό δεν μπορεί να προχωρήσει αυτή η δικασία και να ελεγχθεί διότι τα πάντα ελέγχει ο Άναξ πες για τι πράγματα μιλάμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω ότι δεν ενδιαφέρεται και δεν κάνει διαφοροποίηση και διάκριση ανάμεσα στα κράτη που ε, εφαρμόζουν τους νόμους και το διεθνές δίκαιο και σε κράτη τα οποία καταπατούν καθημερινά το διεθνές δίκαιο και τις ελευθερίες. Έχουμε το περίπτωση του Μαρόκου και την περίπτωση του Ισραήλ. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτή την θλιβερή πρακτική που υπάρχει. Ευχαριστώ δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει και για να δώσουμε περαιτέρω χώρο για την συζήτηση. Και έτσι θα είναι πιο άμεση η επαφή και η συζήτηση με τους συναδέλφους. Ο Δ. Ντε Μοράλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Φυσικά πάντοτε μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συζήτηση, να αμφισβητηθεί το πιο είναι το καταλληλότερο μέσον για τη χρηματοδότηση μια πολιτική. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί κανεί να ισχυριστεί ότι δεν έχουμε πολιτικού στόχου. Στόχο τη ευρωπαϊκή πολιτική ε, γειτονία είναι η ανάπτυξη μιας διαδικασίας σύγκλησης σε όλους τους τομείς που θα συνεπαγόταν για τις χώρες αυτές ε, εγκύτερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα βελτίωση της ευημερίας των πολιτών τους. Και έτσι ε, προσπαθούμε να αξιοποιούμε τις παλιές και δοκιμασμένες μεθόδους που είχαμε δει από τη διαδικασία της διεύρυνσης που όπως γνωρίζετε αποτελεί και το ε, κύριο σημείο αναφοράς. Βεβαίως κάποια σημεία μπορεί να λείπουν λόγω των δεσμευτικών στόχων που προβλέπει η διαδικασία της διεύρυνσης της ένταξης μιας χώρας, εδώ έχουμε μια διαφοροποίηση, αλλά υπάρχουν, υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο και για μας Σαφέστατο είναι ότι δεν, δεν στοχεύουμε μόνο στη βελτίωση της μικροοικονομικής διαχείρισης ή της ικανότητας οικονομικής συναλλαγής με τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά στόχο έχουμε πάνω απ' όλα να ανοίξουν οι κοινωνίες αυτές για τους πολίτες τους, για το δικό τους καλό. Και αυτό το επιδιώκουμε λαμβανωμένων υπόψη των όσων μας λένε οι ίδιες αυτές οι κοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων φυσικά, πρέπει να το σημειώσω και αυτό, και των κυβερνήσεων των κρατών αυτών στόχους όπως διευθορά και δικαιοσύνη δεν αγγίζουμε λέτε. Θα δείτε όμως ότι ε, αν κοιτάξετε τα προγράμματά μας έχουμε πολλούς στόχους σχετικούς με τη δικαιοσύνη και τη διευθορά. και στον εξυγχρονισμό και σε άλλους τομείς. Λέτε επίσης ότι δεν είμαστε αρκετά σαφείς ή δεν μιλάμε αρκετά ανοιχτά όχι, εμείς μιλάμε σε κάθε μας επαφή με αυτούς τους εταίρους για, τη δικαιοσύνη, για, για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δικαιοσύνη και επιδιώκουμε ε, από κοινού μαζί τους να βρούμε τρόπους για την εξασφάλιση αυτής της σύγκλησης, η οποία σύγκληση βεβαίως διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της αναβάθμισης και αυτό το έχουμε πει επίσης και πριν από την εκκίνηση της όλης διαδικασίας, πριν δηλαδή μας υποβάλλουν τις ε, προτάσεις τους με τα σχέδια για την αναβάθμιση ίδιας αυτές τις χώρες. Αυτό το έχουμε επισημάνει σε όλες τις χώρες. Και ως εκ τούτου, όπως και για την Τινησία θα επαναλάβω ότι Έχουμε στη Συμφωνία Συνεργασίας τη ρήτρα των θρηνών δικαιωμάτων και συγκεκριμένα για τη Συρία, όταν εξασφαλίσουμε το νομικό πλαίσιο συνεργασίας με τη Συρία, θα ξεκινήσουμε το διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στη χώρα αυτή. Τι στόχο εξυπηρετεί αυτός ο διάλογος. Ο διάλογος αυτός ε, δεν ε, είναι μόνο θεωρητικός. Έχει σαν στόχο να προαγάγει και αυτές τις αξίες αποτελεσματικά. Η εναλλακτική λύση σε περίπτωση που δεν προχωρεί η συμφωνία σύνδεσης ε, προτιμούμε να μην έχουμε εναλλακτική γιατί θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία και να δίνουμε και χείρα βοηθείας στις ε, δυνάμεις εκείνες της Συρίας που τάσσονται υπέρ της μεταρρύθμισης ε, ταυτόχρονα. Αυτό ρητά το έχουμε δηλώσει όλους μας τους στόχους. Επίση προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε στις προσπάθειές μας την κοινωνία των πολιτών. Έτσι απαντώ καταφατικά στην ερώτησή σας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δημιουργούμε τους όρους δράσης της κοινωνίας των πολιτών. Και πολλές φορές ε, βρισκόμεθα, ξέρετε, ενώπιον του διλήμματος, του κατά πόσον μπορούμε να ε, στηρίζουμε οργανώσεις ε, οι οποίες μπορεί να αποτελέσουν μόνο και μόνο επειδή συνεργάζονται μαζί μας στόχο καταστολής. Αυτό είναι ένα πρόβλημα σοβαρό για μας και μεγάλο δίλημα. Αρκετά συχνό το, συχνά το αντιμετωπίζουμε. Επίσης, θα ήθελα να σημειώσω ως προς την παρατήρηση ότι δεν κάνουμε τίποτε και ότι οι πολιτικές μας, οι στόχοι μας ε, είναι άχρηστοι διότι δεν ε, καταφέρνουμε να κάνουμε τις χώρες αυτές να συμπεριφέρονται όπως θα θέλαμε εμείς, θα λέγω ότι είναι μάλλον άδικη αυτή η κατηγορία. Όσο μας αφορά, όσο αφορά τους στόχους μας, δεν υπάρχει έλλειψη σαφήνειας ή ορατότητας. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να συμμετάσχουμε σε μια διαδικασία κοινωνικής μετάλλαξης μέσω των μεταρρυθμίσεων, η οποία μπορεί να είναι αποτελεσματική επιταχύνοντας και να επιτύχει τους στόχους της, ε, τα ανθρωπινα, την πραγωγή των ανθρώπινων δικαιωμάτων και τη δικαιοσύνη την οποία ε, έχουμε ορίσει ως στόχους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν επισημαίνουμε συνέχεια τους στόχους αυτούς στα διάφορα μέσα και στην ε, πολιτική αυτή της συνεργασίας αλλά και στα οριζόντια μέσα όπως την πολιτική για την προαγωγή των ανθρωπινών δικαιωμάτων και άλλωστε το πράττουμε αυτό συνέχεια και με το διάλογο που αναπτύσσουμε με τις χώρες αυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μοράλ. Πέντε συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Ο χρόνος πιέζει, παρακαλώ, λεπτές παρεμβάσεις. Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ. Λυπάμαι που δεν μπόρεσα να λάβω το λόγο πριν από την παρέμβαση του εκπροσώπου της Κομισιόν, διότι στις 12 ακριβώς πρέπει να φύγω. Θα ήθελα όμως να θέσω κάποιες ερωτήσεις που θα επιθυμούσαν να ληφθούν υπόψη. Πρωτίστως να ευχαριστήσω τον κύριο Μοράλ που ήρθε να μας ενημερώσει σχετικά με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της μεσογειακής πολιτικής. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό που μας έδωσε αυτές τις προφορίες αναφορικά με τα προγράμματα που έχει η Κομισιόν για το στόχο αυτό της mid-term review. Νομίζω ότι είναι μια θετική αξιολόγηση. Θα πρέπει λοιπόν να ευχαριστήσουμε την ε, Κομισιόν για τη συνεργασία της και για την παρουσία της. Ε, παρατηρώ πως ε, αυτό το έργο συμπληρώθηκε και με κάποιες αναλύσεις που έκανε το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να γνωρίζω λοιπόν ποια είναι η αξιολόγηση που κάνει η Ευρωπαϊκή Τροπή αυτών των μελετών, αυτών των αναλύσεων και κατά πώς θα μπορούσαν να τη βοηθήσει στο έργο της. Δεν ε, έχει διανεμηθεί ακόμα το έγγραφο στην Κομισιόν. Ε, ίσως θα πρέπει να τους το διαβιβάσουμε για να δούνε και τα σχόλια που προέκυψαν από το Κοινοβούλιο μετά από αυτή τη μελέτη. Νομίζω ότι το όλο το εγχείρημα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και όπως είπαν και οι συνάδελφοι θα χρειαστεί κατά κάποιο τρόπο να θέσουμε όλες αυτές τις δράσεις ε, ε, σε διμερές επίπεδο σε τέτοιο, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χάσουμε το σύνολο να μην χάσουμε το στόχο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, ε, η, πολιτική μάλλον της, ε, στη Μεσόγειο θα πρέπει να είναι ένα βασικό, μια βασική αρχή της, ε, του μέσου του γειτονίας και όπως είπαν και κάποιοι συνάδελφοι στην πανεβασία τους, αυτό δεν πρέπει να το χάσουμε. Λοιπόν, να θέσω κάποιες ερωτήσεις. το ενδεικτικό πρόγραμμα για την Αίγυπτο, δεδομένου ότι ό,τι αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και υποστήριξη των πολιτικών μεταρρυθμίσεων αποτελούν ε, μόνο το 1,1% από τα 140-150 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν για την ε, δράση αυτή προς την Αίγυπτο από τον ε, προϋπολογισμό μας. Νομίζω ότι μπορεί εύκολα κανείς να κατανοήσει τους λόγους ότι δηλαδή μέσα στο μέσο γειτονίας ε, <clears throat> στο ε, δίνονται μόνο 6 εκατομμύρια ευρώ και εδώ ασκήθηκαν κάποιες κριτικές τις οποίες θα μπορούσα να συμμεριστώ εν, εν τίνη μέτρο. Να πω ότι συμφωνώ για μια φορά με τον κύριο Μέγερ ότι έχουμε συντάξει πάρα πολλέ εκθέσει και θα πρέπει να διευκρινιστεί ο τρόπος εφαρμογής της ρήτρα ε, για τη δημοκρατία στα συμφωνία σύνδεση. <clears throat> Διαπιστώνω με ικανοποίηση την αναφορά στην αποστολή παρατήρησης στον Λίβανο και μια ερώτηση που με ενδιαφέρει πρόεδρο είναι αν τεθεί σε, ενέργεια η συμφωνία σύνδεση με την Συρία αυτό θα σήμαινε κάποιες αλλαγές από πλευράς προϋπολογισμού όχι, και όχι από ποιοτική μόνο σε ό,τι φορά τη στάση και τη σχέση που έχουμε με την χώρα αυτή ο κύριος Πεγιό, εισηγητής της ΑΦΕΤ για την Ένωση του Μητροσυγείου. Τρία λεπτά παρακαλώ. Καταρχάς πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην κάνουμε τη συζήτηση σε σφαλμένη βάση. Πρέπει να στεκόμαστε γερά πάνω και στο σκέλος της οικονομικής συνεργασίας και στο σκέλος των ε, ανθρωπινών δικαιωμάτων και των ε, ε, δημοκρατικών προϋποθέσεων Αυτά είναι απαραίτητα στοιχεία για μας, δεν μπορούμε να λησμονούμε το ένα και το άλλο. Και ο κύριος Αλαφράγκα είπε, όπως η κυρία Φλότρο, ότι πρέπει να στηριζόμαστε πάνω στα δύο σκέλη, αλλά η ισορροπία δεν είναι η βέλτιστη. Έχουμε ίσως επιβάλει ένα μοντέλο με την συμφωνία ένα μοντέλο σε δύο σκέλη, αλλά ταυτόχρονα συμφωνώ και εγώ με του συναδέλφους ότι πρέπει να επιμείνουμε ιδιαίτερα ώστε να αποκαταστήσουμε τη σημασία κάποιων από, των προϋποθέσεων, από τις προϋποθέσεις που θεωρούμε πολύ σημαντικέ. Και επίση, ιδιαίτερα εμεί, ε, το Κοινοβούλιο δηλαδή, θέλουμε και επιμένουμε να αναπτυχθεί η αποτελεσματικότητα αυτής της πολιτικής γειτονίας βεβαίως, αλλά να αναπτυχθούν ταυτόχρονα και η συνεργασία μας και οι δεσμοί μας με τον Νότο μεγάλη σημασία και αυτός ο στόχος. Έτσι λοιπόν έρχομαι στο εξή. Γιατί ήθελα κάποιε διευκρινήσει Από το 2007 έχουμε την Ένωση για τη Μεσόγειο. Και ύστερα από και παρά μάλλον τις προσπάθειες ή με τις προσπάθειες που κατεβλήθησαν φαίνεται να ε, προχωρεί η υπόθεση αυτή σιγά σιγά και θα ήθελα να μάθω τι είδους δεδομένα έχουμε για την πορεία αυτή της Ένωσης για Μεσόγειο, τα έγγραφα στρατηγικής 2007-2013 και μέχρι τίνου σημείου, θα ήθελα να πείτε, βλέπετε κάποια δυνατότητα για την Επιτροπή, γιατί υπήρξαν ανησυχίες ανησυχίες να προωθήσει τη συμπληρωματικότητα της Ένωσης για τη Μεσόγειο με τα νέα ενδεικτικά, εθνικά ενδεικτικά προγράμματα που προετοιμάζονται για τον ορίζοντα το 2011-2013. Τι όραμα έχετε λοιπόν ως προς την ενσωμάτωση, το συντονισμό αυτών των πολιτικών γειτονίας. Ευχαριστώ. Μπιναράμπ Ατού, τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίχθηκε στη βούληση να μην ξαναζήσουν οι λαοί της τα δεινά του πολέμου. Και τώρα αυτή τη βασική βούληση πρέπει και εμείς να την αναπτύξουμε σε μια, μια βάση ειρήνης και σταθερότητας έναντι των εταίρων μας, έτσι ώστε να ξεφύγουν από το φαύλο δολοφονικό κύκλο της βίας. Πρέπει λοιπόν πρώτον να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της ε, σκληρής επικιστικής πολιτικής του Ισραήλ. Δεύτερον, να στρώσουμε ένα τέλος στις τρομοκρατικές ενέργειες που τους, το θάνατο και τρίτον, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που προσπαθούν από την νότια όχθη να περάσουν, διακινδυνεύοντας και τη ζωή τους στη βόρεια όχθη της Μεσογείου, του Χάρακα. Εάν δεν αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά, θα μπορέσουμε να καταφέρουμε τίποτα. Οι συμφωνίες σύνδεσης και οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να μας επιτρέπουν τις προϋποθέσεις αυτές ε, να τις ε, υλοποιήσουμε και να δώσουμε λύση στα φαινόμενα αυτά. Οι Χάραγκα, λοιπόν, αυτοί οι νέοι μετανάστε, ε, έχουν ένα παρουσιάζουν ένα πρόβλημα διτό. Οι χώρες της Νότιας Όχθης Μεσογείου και ιδιαίτερα του Μαγκρέπ παρουσιάζουν ε, συνθήκες ζωής ικανοποιητικές για τις κοινωνίες τους, ανοιχτές κοινωνίες με δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, πλουραλισμό, ελευθερία της ε, έκφρασης της γνώμης, της πολιτικής ε, βούλησης. Αυτός θα πρέπει να είναι ένας στόχος για μας. Δεύτερον, θα πρέπει η πολιτική που θα αναπτύξουμε να μην οδηγήσει σε ανάπτυξη ανισοτήτων για εκείνους που μπορούν να περάσουν, εκείνους που δεν μπορούν να περάσουν στη βόρεια όχθη της Μεσογείου. Η νότια όχθη είναι το όριο, η μεθόριος και ιδιαίτερα το σύμβολο του τύπου των σχέσεων που θέλουμε να αναπτύξουμε εμείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον υπόλοιπο κόσμο και όχι μόνο με την νότια όχθη του Μεσογείου. Ευχαριστώ. Πανσιέρη. Πρόεδρος της Αντιπροσωπής για σχέση με το Μαγκρέπ. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπάρχει κάτι γενικότερο, εντάξει, θεωρώντας θετική την προσέγγιση από πλευρά Κομισιόν, πιστεύω πως χρειάζεται να βάλουμε λίγο πιο ψηλά τον πύχη για τον στρατηγικό ρόλο που η περιοχή μπορεί να διαδραματίσει γενικότερα. Και θα ήθελα η Κομισιόν να κατανοήσει πως ε, απαιτείται μια μεγαλύτερη όθηση ε, αυτό θα μας βοηθήσει να βρούμε κάποιες μάλτες ισορροπίες στην πολιτική γειτονία. Τώρα, οι παρατηρήσεις μου έχουν ως εξής στην πολιτική γειτονία θα πρέπει να υπερισχύσουν δύο θέσεις που αλληλοσυγκρούονται. Ένας υπερβολικός ρεαλισμός, ο οποίος ε, βασίζεται στο ότι οι διμερείς συμφωνίες και όχι μόνο γίνονται και αφορούν αποκλειστικά την οικονομική πτυχή της ανάπτυξης και να έχουμε ως μοναδικό σημείο αναφοράς το ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι σημαντικότατο, είναι πολύ σημαντική η δημοκρατική ρήτρα με μια στάση μάλλον υπερβολική που πολλές φορές και στις συζητήσεις μας ακόμα απέναντι σε μια παραβίαση ε, ετοιμαζόμαστε να διακόψουμε τις διπλωματικές σχέσεις με κάποια κράτη. Η ισορροπία πετυχάνεται, όπως είπε και ο συνάδελφος Πεγιών, εάν δράσουμε και στις, στα δύο σκέλη του ζητήματος, στην δημοκρατική ε, στην ανάπτυξη αλλά και στην ε, δημοκρατία και τις δημοκρατικές εξελίξεις. Αυτό πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο του γενικού διαλόγου της Λεκάνης Μεσογείου αλλά και στις διμερές επίπεδο και καταλήγω ζητώντας από την Κομισιόν να σκεφτούν κάποια ζητήματα, διότι εγώ βλέπω εδώ κάτι που αλληλοσυγκρούεται όπως η, θέση της Ευρώπης και η προσέγγιση της στην περιοχή και οι δράσεις των επιμέρους κρατών που σε διμερές επίπεδο πολλές φορές ε, με την θέση της Ευρώπης. Θα ήθελα να γνωρίζω λοιπόν και ρωτώ την Κομισιόν πώς προτίθεστε να δράσετε ανάμεσα στις ε, θέσεις ε, των επιμέρους κρατών μελών, ειδικά των χωρών της Μεσογείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Κιλ Νίλσεν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ό,τι αφορά την τήρηση του διεθνούς δικαίου και ειδικά στο πλαίσιο των σχέσεων με το Ισραήλ, λαμβάνοντας κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα, να μιλήσω για την οικοδόμηση και εκμετάλλευση μιας υπογείου ε, σύνδοτρομου που θα ενώνει τις ε, επικισμούς και τα παράνομους κατεχόμενα εδάφη από το 67 και τη μιας γαλλικής επιχείρησης η οποία ανέλαβε αυτό το πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται ήδη. Τώρα το ζήτημα του ύδατος, η τεχνολογία του ύδατος θα πρέπει να επωφελεί προς όφελος ε, της Ευρώπης. Αλλά τι γίνεται με το δικαίωμα στο νερό. Θα σας πενθυμίζω ότι τον Οκτώβριο η Amnesty International εξέδωσε μια έκθεση πολύ σημαντική για τον περιορισμό σε ό,τι φορά την πρόσβαση του ύδατος στις κατεχόμενες περιοχές της Παλαιστίνης. Λοιπόν, είναι, το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Είχα θέσει την ερώτηση γραπτό στην Κομισιόν και κάποια στιγμή θα μου απαντήσει τι μέτρα και τι μηχανισμούς ελέγχου προβλέπει ώστε τα αγροτικά προϊόντα τα οποία εισάγονται στην Ευρώπη να μην προέρχονται από εκμεταλλεύσεις ε, παλαιστινιακές που βρίσκονται υποκατοχή. Και ένα άλλο θέμα, το θέμα της δημοκρατίας, της Ισραηλινής δημοκρατίας, τι έγινε με τους 35 νόμους που στο Ισραήλ δίνουν προτεραιότητα στους ε, ε, Εβραίου και, τι, και αποτελούν διάκριση πάνω των Παλαιστινίων και τι γίνεται με τους ειρηνιστές ε, Ισραηλινούς, είτε είναι Ισραηλίτες είτε Άραβες, οι οποίοι συνέρχονται κάθε εβδομάδα στο Σεκ Ζαρά για να ε, διαμαρτυρηθούν κατά της ε, <clears throat> απομάκρυνσης ε, κατοίκων στην ε, Ανατολική Ιερουσαλήμ. Θα ήθελα λοιπόν να Κώστος ότι ε, πρέπει επίσης να ακούσουμε την κοινωνία των πολιτών. Είναι σημαντικό αυτό και σα καλώ να έρθετε απόψε το βράδυ σε μια συνάντηση που οργανώνουν Στάρφη και εγώ. Προσκαλέσαμε μέλη μιας Ισραηλινο-Παλαιστινικής οργάνωσης Combat for Peace Εξ αυτών ε, βρίσκονται στην αίθουσα και θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να ακούσετε μια Ισραηλινή γυναίκα η οποία νέα, η οποία υπηρέτησε στον Ισραηλινό στρατό και τώρα είναι, ε, συμμετέχει σε αυτήν την δράση για την ειρήνη, να μας ε, πει δηλαδή τι είναι αυτό που περιμένουν από την Ευρώπη. Δηλαδή θεωρούν ότι το καθήκον μας είναι να βοηθήσουμε το Ισραήλ να γίνει μια δημοκρατική χώρα, να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, να θέσει τέλος στο φιλετιστικό καθεστώς, το Apartheid και μας λέει ότι περιμένει και προσδοκά πολλά από την Ευρώπη ακριβώς σε αυτό το ζήτημα της πραγματικής δικαιοσύνης που θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Κίρ Νίλσεν για τα τελικά σχόλια. Ο κύριος Ντεμοράλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς να πω ότι δεν πιστεύουμε. σε καμία περίπτωση ότι υπάρχει έλλειψη ευαισθησίας. Εδώ υπάρχουν διλήμματα τα οποία θα πρέπει να αποφασιστούν. Καταλαβαίνω τι λέμε, ότι παρά την ε, ανάγκη να είμαστε ρεαλιστικοί, πρέπει παράλληλα να είμαστε και φιλόδοξοι σε ό,τι αφορά την προώθηση των αξιών μας στους εταίρους μας. Και νομίζω ότι το σημειώνουμε με το σωστό τρόπο το σημείο αυτό. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί την βάση των ενεργειών μας. Ίσως όμως η έκκληση να σημαίνει ότι θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε πιο έντονα. Ίσως θα πρέπει να το εξετάσουμε. Ωστόσο, αν, ε, αν εφαρμόζαμε κάποιον πύχη περιοριστικό, ο οποίος θα έπρεπε να επιτευχθεί για τη συνεργασία μας με τους ε, εταίρους μας, κάποιους όρους για παράδειγμα, για την εισδοχή στο Συμβούλιο της Ευρώπης, μπορεί τελικά να καταλήγαμε σε μια κατάσταση που δεν συνεργόμαστε με κανέναν από τους εταίρους μας. Και αυτό θα ήταν ιδιαίτερα προβληματικό. Πιστεύουμε και ελπίζουμε και εσείς το ίδιο να πιστεύετε ότι ο τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών είναι να προωθήσουμε τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που τελικά θα βοηθήσουν τις χώρες να υιοθετήσουν τα απαραίτητα μέτρα και θα τις φέρουν πιο κοντά στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του διαλόγου ο οποίος θα πρέπει φυσικά να λάβει υπόψη και τις διαφορές της πολιτισμικές, όχι μόνο τις πολιτικές. Δεν θα ήθελα να περιοριστώ όμως σε γενικά σχόλια, γιατί έγιναν και κάποιες πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις. Για παράδειγμα, για την Αίγυπτο, κατά πόσο το ποσό που δαπανάμε για την υποστήριξη των πολιτικών μεταρρυθμίσεων είναι περιορισμένο, το οποίο μπορεί να εξηγηθεί, επειδή δεν μιλάμε για την παροχή υπηρεσιών για εκατομμύρια πολιτών, όχι, μιλάμε για πράγματα που μπορούν να επιτευχθούν με μικρές οργανώσεις. Μιλάμε για σχέδια τα οποία μπορούν να καταστηθούν, τα οποία δεν συνεπάγονται τεράστια έξοδα και τα χρήματα αυτά που τα δαπανώνται μπορεί να αρκούν αν χρησιμοποιηθούν με σωστό τρόπο. Δεν μιλάμε για χρηματοδότηση υποδομών, που είναι πολύ πιο δαπανηρή, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της ρήτρας της δημοκρατικής για τις συμφωνίες αυτές. Νομίζω ότι δίκιο έχει ο κύριος Σαλαφράγκα που λέει ότι δεν υπάρχει ενιαία και ομοιόμορφη θεώρωση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί μια τέτοια ρήτρα δεν έχω να πω κάτι παραπάνω στις χώρες που έχουν συμφωνίες εταιρικής σχέσης. Δεν γνωρίζω να έχει γίνει οποιαδήποτε αίτηση ποτέ για αναστολή τέτοια συμφωνίας. Θα είναι σημαντικό σε κάποια φάση, αλλά όχι στα πλαίσια του εγχειρήματο αυτού, να δούμε ποια θα είναι τα κριτήρια για την χρήση αυτού του εργαλείου. Όπως σας είπα όμως, πρόκειται για μια πολύ περιορισμένη άσκηση δεν μπορεί να λύσει ένα τόσο σημαντικό και μεγάλο πρόβλημα για το κατά πόσο θα υπάρχουν ε, αλλαγές στη σχέση μας με τη Συρία αν υπογράψουμε τη συμφωνία ασφαλώς. Πολλοί τομεί συνεργασίας θα ανοίξουν και θα πρέπει να αναπτυχθούν μέσω υποεπιτροπών όπως γίνεται και με άλλες χώρες και προσπαθούμε να προγραμματιστούμε να κάνουμε τον προγραμματισμό μας σε περίπτωση υπογραφής της συνθήκης για να έχουμε περισσότερες δυνατότητες για την Ένωση για τη Μεσόγειο. Φαίνεται ότι υπάρχουν προοπτικές πλέον. Θα εγκριθεί το καθεστώς της γραμματείας και θα λειτουργήσουν οι σχετικοί θεσμοί. Θα ήθελα να πω ότι εμείς εντάσσουμε τον προγραμματισμό μας τα όσα έχουν γίνει για την Ένωση για την Μεσόγειο. Τα προγράμματα που εγκρίθηκαν στο Παρίσι πρέπει να πούμε ότι οι πιο σημαντικές συμβολές ήταν από τομείς που ήδη υπήρχε εξέλιξη. Τέσσερις ε, από τους έξι τομείς που προτάθηκαν ήταν τομείς που ήδη είχαν τεθεί σε εφαρμογή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας είπα ότι έχουμε εγκρίνει 70 εκατομμύρια ήδη για την περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτό θα αυξηθεί σε 96 εκατομμύρια για την περίοδο 2011-2013. Και αυτό θα μας επιτρέψει περισσότερα τέτοια προγράμματα συνεργασίας. Ωστόσο, η φιλοδοξία των προγραμμάτων για την Ένωση για τη Μεσόγειο φυσικά ξεπερνά κατά πολύ αυτά που μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε στο περιφερειακό επίπεδο. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν χρηματοοικονομικά εργαλεία για το EID, αλλά και για τους διεθνείς θεσμούς. Και πέραν τούτου θα πρέπει να προσελκύσει το ενδιαφέρον του ιδιωτικού τομέα. Και αυτό θα πρέπει να αποτελέσει μία από τις βασικές ε, εργασίες, τα βασικά καθήκοντα της γραμματείας να συγκεντρώσει όλες τις χρηματοδοτικές πηγές για τις μεγάλες προτεραιότητες που έχουν αποφασιστεί στο πλαίσιο της ε, Ένωσης για τη Μεσόγειο. Συμφωνώ ότι για να επιληθούν τα προβλήματα που σχετίζονται με την μετανάστευση θα είναι να εργαστούμε προς την κατεύθυνση μια πιο ανοιχτής κοινωνίας και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία. Το είπα και εισαγωγικά, το επαναλαμβάνω και τώρα, για να περιορίσουμε και μέσω του διαλόγου τον αριθμό των ανθρώπων που χάνονται, που πεθαίνουν λόγω της, ε, του συστήματος αυτού. Πώς θα συνδυαστεί η απαραίτητη αντίδραση για κάθε μεμονωμένη χώρα με τη γενική μας πολιτική. Όπως σας είπα, αυτό θα πρέπει να το κοιτάξουμε εξατομικευμένα για κάθε χώρα. Και πώς θα γίνει αυτό. Θα πρέπει να υπάρχουν διάφορα σχέδια δράσης, ενδεικτικά προγράμματα για κάθε χώρα. Κατά δεύτερον, να είναι καλές οι δομές του διαλόγου για να, μπορέσουμε, να μπορούμε να συζητάμε τα προβλήματα όπου αυτά ανακύπτουν είτε όταν αφορούν ε, τις δομές της συμφωνίας ε, εταιρική σχέσης, είτε όχι. Και φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παράδοση ανταπόκρισης σε ό,τι σημαίνει στον κόσμο, στα τεκτενόμενα, μέσω δηλώσεων, διακηρύξεων, διαβημάτων. Δυστυχώς τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας δεν είναι άμεσης ε, ανταπόκρισης. Μιλάμε πιο πολύ για εργαλεία μεσοπρόθεσμων αλλαγών. Έχουμε σχετικά μέσα, αλλά δεν εντάσσονται, όπως είπατε, στο πλαίσιο του παρόντος εγχειρήματος, όπως για παράδειγμα το μέσο για την σταθερότητα, για τους μικρατικούς φορείς και όλα αυτά δεν είναι όμως ιδιαίτερα ευέλικτα ούτε αυτά τα εργαλεία ούτε πολύ ταχείας αντίδρασης. Έτσι έχουν όμως τα πράγματα. Τώρα, δεν προσπαθώ να παρακάμψω τα συγκεκριμένα προβλήματα που αναφέρθηκαν σε ό,τι αφορά τη σύγκρουση στη Γάζα. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο αντιμετώπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητώντας από το Ισραήλ να περιορίσει αλλά και τις δράσεις του και ενισχύοντας ε, τους πληθυσμούς που ε, πλήττονταν. Θεωρούμε ότι ο καλύτερος τρόπος για την επίλυση των προβλημάτων είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την ειρήνη. Ένας από τους πυλώνες είναι η οικοδόμηση του Παλαιστινιακού κράτους και προσπαθούμε να βοηθήσουμε την Παλαιστινιακή Αρχή για την οικοδόμηση αυτού του κράτους ακολουθώντας τις γραμμές της ε, Παλαιστινιακής Αρχής. Δυστυχώς το θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε να επιλύσουμε τα πολύ σοβαρά ζητήματα που μαστίζουν την περιοχή. Είτε πρόκειται για την οικονομική κατάσταση του Παλαιστινιακού λαού και στη Γάζα, που δεν εξαρτάται μόνο από τους επικισμούς αλλά και από άλλους παράγοντες, είτε την κατάσταση στην Ανατολική Ιερουσαλήμ καταβάλουμε προσπάθειες σε πολιτικό, διπλωματικό επίπεδο, επίπεδο συνδρομής, σχέδια δράσης, διάλογο, ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να συνδράμουμε στην ειρηνευτική διαδικασία. Νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε τον κύριο Μοράλ. Μια τον επικοδομητικό διάλογο που είχαμε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που συνεισέφεραν σημαντικά σε αυτόν τον διάλογο. Στους προσεχείς μήνες θα υπάρξουν εξελίξεις και από πλευράς κομισιών ακούσαμε ότι θέλει να ενισχύσει την ε, οικονομική της συνεισφορά. Σας ευχαριστώ όλες και όλους. Θα επαναληφθεί η συνεδρίασή μας στις 15.00 ε, με την Προεδρία του Συνέδελφου Προβέρα, όπου θα εξετάσουμε τις ε, χώρες της Ανατολικής και δει την κατάσταση στη Γεωργία.